So, liebe Kolleginnen und Kollegen, guten Tag und herzlich willkommen zu der Ausschusssitzung. Ich... Ξεκινάει η συνεδρίασή μας, αγαπητοί συνάδελφοι. Καλώς ήρθατε όλοι. Στο σημείο 1 της ημερήσιας διάταξης έχουμε την έγκριση της διάταξης. Θα υπάρξει μια αλλαγή η ανταλλαγή απόψεων με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων θα αναβληθεί γιατί το άτομο επαφή η Dagmar Μπέρεντ, είναι άρρωστη και δεν μπορεί να παραβρεθεί στην συνεδρίαση σήμερα. Έχουμε λοιπόν ένα κενό. Επειδή το επόμενο σημείο στην εμερήσια διάταξη αφορά τα επικίνδυνα χημικά προϊόντα. Και ο κύριος Νταν Γιώργενσεν ε, θα έρθει στις 5 μόλις για να συζητήσουμε. Άρα, όταν θα τελειώσουμε και το σημείο 4, θα κάνουμε ένα διάλειμμα μέχρι τις 5 και μετά θα έρθει και η Επίτροπος Χέρικαρτ. Ωραία, λοιπόν. Να περάσουμε τώρα στο σημείο 2 της ημερήσιας διάταξης. Θα μάθατε ίσως όλοι ότι σε ό,τι αφορά την εκτίμηση για τις εκπομπέ του διοξιδίου του άνθρακα και μια ε, έκθεση και είχαμε πραγματικά εκπομπή ρεκόρ τέτοιων αερίων. Αυτό πραγματικά είναι δυσάρεστο γιατί δεν σημειώνουμε πρόεδρο. Μην σας πω ότι σημειώνουμε και ε, επαναχώρηση. 6% πιο πολλά αέρια το 2010 από το 2009. Αυτό σίγουρα θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε και ως όπλο σε ό,τι αφορά το ψήφισμα για τον Τέρμπαν που θα ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα. Ύστερα είχαμε την σύνοδο του G20 που έπρεπε να ασχοληθεί και με θέματα περιβάλλοντος, αλλά ασφαλώς δεν μπόρεσε να φτάσει στο θέμα αυτό λόγω των, ε, της χρηματοπιστωτικής ε, και της κρίσης του ευρώ. Αναφέρονται ωστόσο δύο παράγραφοι από τους πλέον ισχυρούς του κόσμου και το G20 επιβεβαιώνει ότι οι επιδοτήσεις για ορεικτά καύσιμα πραγματικά πρέπει να λάβουν ένα τέλος στην τρέχουσα δεκαετία. Και έτσι σε ό,τι αφορά τον Τέρμπαν, κατά τα άλλα, μόνο αεροστρολογίες έχουμε. Γενικούρες, γιατί δυστυχώς δεν κατάφεραν να ασχοληθούμε το θέμα αυτό. Περνάμε τώρα στην έγκριση των πρακτικών 13-14 Ιουλίου του 12 Σεπτεμβρίου, 26 Σεπτεμβρίου, 3 έως 5 Οκτωβρίου. Ως συνήθως, αν δεν ε, έχουν διατυπωθεί αντιρρήσεις μέχρι το τέλος της συνεδρίας, θεωρούνται εγκεκριμένα τα πρακτικά. Και τώρα ξεκινάμε. Στο σημείο 4. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό να καλωσορίσω την ε, διευθύντρια, την εκτελεστική διευθύντρια της ΕΦΣΑ τη, από την Πάρμα, την κυρία Καθρίν Βεσλέν Λενέλ και την ε, ομάδα της, κυρία Ζεσλέν Λανέλ. Πάντα είμαστε ευτυχείς όταν έρχεστε στην Επιτροπή μας. Χαίρετε λοιπόν η Επιτροπή που βρίσκεστε εδώ, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική η υπηρεσία η ΕΦΣΑ ασχολείται με θέματα τα οποία μπορεί να είναι πολύ αμφιλεγόμενα. Και σήμερα έχουμε την ετήσια παρουσίαση του προγράμματος εργασίας για, το, για την ΕΦΣΑ. Άρα τα μέλη της ομάδας, τα μέλη της Επιτροπής ανυπομονούν να ακούσουν τι έχετε να μας πείτε και γι' αυτό σας δίνω ευθύ αμέσως το λόγο. Καλώς ορίσατε λοιπόν. Dear Chair, Honorable members. Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, ε, Χαίρομαι ιδιαίτερος ε, που ετησίως έχω την ευκαιρία να μιλώ ενώπιον του Κοινοβουλίου. Οι εργασίε μα, με στόχο την προστασία των πολιτών έχουν ιδιαίτερη σημασία και είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονε για τη συνεργασία που έχουμε με το Κοινοβούλιο. Τα τελευταία χρόνια έχουμε διαβουλευτεί για βασικά ζητήματα και το ενδιαφέρον που δείχνεται για τις εργασίες μα το εκτιμούμε ιδιαίτερο. Θα ήθελα σήμερα να σας ενημερώσω για τι εργασίε μα το έργο μα, σε τρει ε, βασικού τομεί ε, που έχουν πολύ σοβαρέ επιπτώσει για την ε, υγεία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα χημικά, στα τρόφιμα, την διατροφή και τις ε, χημικές ουσίες ε, μέσα στα τρόφιμα καθώς ε, και τις τροφιμογενείς ασθένειες. Στη συνέχεια θα σας μιλήσω για τις στρατηγικές εξελίξεις στον ΕΦΣΑ. Τα κρούσματα ή κόλλη στη Γερμανία και την Γαλλία νωρίτερα φέτος Μα έδειξαν πέραν κάθε αμφιβολία στη σημασία τη ελέγχου των οσογόνων μικροοργανισμών, η τραγική έκβαση δηλαδή μέχρι 50 νεκροί, χιλιάδε που ασθενούν και εκατοντάδε που έχουν πλέον μόνιμε αναπηρίε μα υπενθυμίζουν ε, τι ζημιέ που μπορούν να προκαλέσουν οι τροφιμογενεί νόσοι, οι ζωονόσοι μεταβιβάζονται από τα ζώα προ του ανθρώπου ε, και ε, συμπεριλαμβάνουν του μικροοργανισμού στην Ευρώπη έχουν το μεγαλύτερο μεγαλύτερο επιπελασμό και είναι τροφιμογενείς όπως η σαλμονέρα και το καμπυλοβακτηρίδιο. Είναι σημαντική απειλή. Πάνω από 320.000 κρούσματα αναφέρονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε χρόνο, αναγνωρίζοντας τη σημασία που έχουν για την δημόσια υγεία την περασμένη εβδομάδα η Αντιπρόεδρος ε, κυρία Ροτ δύο διοργάνωσε και προείδρευσε σε ένα σεμινάριο εδώ στο Κοινοβούλιο. Συνδιοργανώθηκε το σεμινάριο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κέντρο, ε, Κέντρο Ελέγχου των Νόσων, το ΕΚΠΕΜ, Σημειώθηκε ιδιαίτερη πρόοδο στην χαρτογράφηση τη πρόοδου καταπολέμηση τη ασθένεια αυτή στην Ευρώπη ε, και συζητήθηκε το θέμα του ελέγχου των ζωονόσων. Ε, στην περίπτωση τη Αλμονέλα ε, είχαμε μείωση κατά το ίμιση των κρουσμάτων στου ανθρώπου για την πενταετή περίοδο μέχρι το 2009 και νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό, κυρίω υπό το φω των παγκοσμίων τάσεων. Το έργο τη ΕΦΣΑ έπαιξε κύριο ρόλο για την επίτευξη αυτού του στόχου και φυσικά είμαι προτιθέμεθα να υποστηρίξουμε ε, κάθε εθνική και ευρωπαϊκή προσπάθεια. Ε, τα ζωικά μας κεφάλαια είναι ε, οι βασικές αιστείες ε, μολυσεών από ζωνόσους ε, και γι' αυτό ε, λάβαμε μια ευρύτατη εντολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2010 για να συγκροτήσουμε μια επιστημονική βάση για τον εξχρονισμό του ελέγχου του κρέατος στην Ευρώπη. Εντοπίζουμε συγκεκριμένους βιολογικούς κινδύνους συμπεριλαμβανομένης και της αλμονέλας και αναδεικνύουμε νόσους όπως η σαλμονέλα σε προτεραιότητες κυρίως για την επιθεώρηση του χειρίου, πρέβατος, του χειρίου συγγνώμη, κρέατος ε, στα σφαγεία. Ε, προτείνουμε νέες μεθόδους ε, ελέγχου. Επίσης, ε, θέλουμε να προωθήσουμε την πρόορη διάγνωση των βιολογικών κινδύνων, καθώς και την εισαγωγή ένας συνολικού πλαισίου για τα σφάγια των χείρων και στρατηγικές που θα βασίζονται στην ανάλυση του κινδύλου. Μέχρι τα μέσα του 2013 θα έχουμε δημοσιεύσει έξι γνωμοδοτήσεις με στόχο να ελέγχουμε καλύτερα τις μολυματικές ουσίες βιολογικού ή ε, τις βιολογικές και χημικές ε, μολυσματικές ουσίες ε, στην αλυσίδα του κρέατος στην Ευρώπη. Τα κρούσματα του E. καταδεικνύουν ότι όταν είμαστε καλά προετοιμασμένοι για τις κρίσεις μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πιο αποτελεσματικά τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Ε, από τότε που ξέσπασε η κρίση, τον Μάιο και τον Ιούνιο, έχουμε εκδώσει έξι διαφορετικές νομοδοτήσεις και εκθέσεις. Ε, αποκινούμε το ΕΚΠΕ και άλλους ε, οργανισμούς ε, γνωμόνων στα κράτη-μέλη. Επίσης, κατόπιν ετοίματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Γερμανικών Αρχών, αντιπροσωπεία της ΕΦΣΑ, ε, τεχνική αρρωγή για την αντιμετώπιση της ε, κρίσης. Όταν προέκυψαν κρούσματα και στη Γαλλία, συντονίσαμε μια task force, ώστε να εξετάσουμε την πιθανή στενή σχέση που υπάρχει ανάμεσα ε, στις αιστείες ε, λόγω των ε, Ε, λόγω, τους ε, σπόρους, ε, λόγω των σπόρων που εισάχθηκαν από την Αίγυπτο στην Γερμανία. Τα τελευταία χρόνια έχουμε προοδεύσει πολύ ως προς την ανάλυση των δεδομένων, την παρακολούθηση των στατιστικών στοιχείων για τους ναδιόμενους κινδύνους και έτσι η Ευρώπη μπόρεσε να δώσει μια πιο αποτελεσματική απάντηση για τους σπόρους τριγωνέλας. Σε σχέση λοιπόν με την επικοινωνιακή μας πολιτική για τη του κινδύνου. Ε, έχουμε και το Συμβουλευτικό Φόρουμ και τι σχετικέ κατευθυντήριε γραμμέ που μα βοηθούν για την μετώπιση των ευρωπαϊκών ε, κρίσεων. Και σε σχέση με τη θεματική μα προσέγγιση, όπω ανακοινώνεται στη στρατηγική μα ε, για την ανακοίνωση στοιχείων για την περίοδο 2010-2013, στην ιστοσελίδα μα θα βρείτε πλήρε πληροφορίε για τι ζωονόσου. Τώρα, σχετικά με τα, τις χημικές ουσίες στα τρόφιμα. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία στην κοινή γνώμη, όπω φαίνεται από πρόσφατε δημοσκοπήσει ε, του Ευρωβαρόμετρου σχετικά με τι ε, χημικέ ουσίε ε, στα τρόφιμα και τα υπολείμματα από ζυζανιοκτώνα. Έχουμε αρχίσει την ετήσια συλλογή των ρηπογόνων ουσιών, ουσιών ανακράτος μέλος και έχουμε ελέγξει τα ε, συστήματα ελέγχου. Έχουμε ασχοληθεί με υπολείμματα φαρμάκων, ε, με ε, μόνιμους οργανικούς ρήπους όπως οι διοξίνες και τα πολυχλωριωμένα διφενήλια καθώς και τα υπολείμματα των ζυζανιοκτώνων ε, που συμπεριλαμβάνουν ε, ε, ουσίες όπως οι αφλατοξίνες, τα φουράνια και το ακριλαμίδιο που χρησιμοποιούνται κατά την επεξεργασία των τροφών. Επίση, ενισχύουμε την αξιοπιστία των δεδομένων και συνεχίζουμε στενή συνεργασία με τον ΠΟΗ και τον ΦΑΟ. Μέσα από αυτέ τι μελέτε εκτιμούμε το επίπεδο των ρηπογών ουσιών μέσα στι τροφέ, καθώ καταναλώνεται και το, την τροφή ε, την έχουμε προετοιμάσει φυσικά προτού διεξάγουμε οποιαδήποτε ανάλυση. Ε, βάσει μια νομοθεσία ε, που άρχισε να υλοποιείται το 2008, τα κράτη-μέλη διεξαγάγουν ετήσια προγράμματα παρακολούθηση ε, για τα υπολείμματα των ζυζανιοκτώνων και αναφέρουν τα αποτελέσματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην ΕΦΣΑ. Αύριο θα δημοσιεύσουμε την τρίτη ετήσια έκθεση για τα υπολείμματα αυτό, κάνοντα μια επισκόπηση των υπολείμματων που έχουν εντοπιστεί σε τρόφιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το 2009. Τα πορίσματα είναι ενθαρρυντικά και μα δείχνουν ότι ότι η συμμόρφωση συνεχίζει να αυξάνεται. Τα υπολείμματα από πάνω από 800 οκτώνα ε, ήταν εντός ε, των ε, ορίων που συστήνονται σε 98% από τις 68.000 από τις 68.000 δειγματοληπτικούς ελέγχους που έγιναν. Επίσης δείχνει η έκθεση ότι 61,4% των δειγμάτων ήταν ελεύθερα από τέτοια υπολείμματα που μπορούν να μετρηθούν καθώς και από τα δείγματα προκύπτει ε, ότι ε, το ποσοστό ε, που υπερβαίνει τις μέγιστες συνιστούμενες ποσότητες έχει πέσει από το 4,4% στο 1,4% σε σχέση με το 2006. Από πλευράς αξιολόγησης κινδύνου και τροφικής πλευράς είναι σημαντικό να ξέρουμε τι, τι τρώνε οι Ευρωπαίοι και να γνωρίζουν επίσης και τη σύνθεση των τροφίμων. Τα τελευταία χρόνια έχουν έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος σε σχέση με την ακρίβεια των δεδομένων που είναι διαθέσιμα για την ΕΦΣΑ ω προ την κατανάλωση τροφίμων των ελληνικών των παιδιών και των ηλικιωμένων. Επίση, ολοκληρώσαμε το έργο μα σε σχέση με την βάση δεδομένων που περιέχει πολλέ λεπτομέρειε για τι ημερήσιε τροφικέ συνήθειε σε περίπου 70.000 ατόμων σε ολόκληρη την Ευρώπη με συνεισφορέ ω προ τα δεδομένα από 22 κράτη-μέλη και που έχουν συλλεχθεί από 32 διαφορετικέ εθνικέ τροφικέ ε, επιστημονικέ επισητιστικές μελέτες, ε, ε, καρδιακιακές επαθήσεις, ε, καρκίνη διαβήτης και χρονικές, χρόνιες αναπνευστικές ενώσεις. Επίσης, οι μη μεταδιδόμενες ασθένειες, οι λεγόμενες, είναι υπεύθυνε για τους τρεις από τους πέντε θανάτους σε παγκόσμια κλίμακα και αυτές οι νόσοι οφείλονται σε ατυχείς διατροφικές επιλογές, έλλειψη σωματικής άσκησης και άλλους παράγοντες σχετίζονται με τον τρόπο ζωή μα. Ένα από τα βασικά προληπτικά μέτρα είναι η παροχή πληροφοριών, η παιδεία ουσιαστικά σε σχέση με το τι συνιστά ε, μια υγιεινή διατροφή. Ε, πέρα από τι βάσει δεδομένων για τι κατα... για τις καταναλώσει τροφίμων, εργαζόμαστε επίση ε, για την εκπόνηση των διατροφικών πολιτικών και για τον προσδιορισμό στόχων για τη δημόσια υγεία που σχετίζονται με την διατροφή καταστροφή του πληθυσμού. Τον περασμένο Ιούλιο ε, περάσαμε και ένα ορόσημο γιατί δημοσιεύσαμε την τελική ε, σειρά των ε, αξιολογήσεων σχετικά με την δημόσια υγεία και είδαμε ότι ήταν το απόγειο της ε, τριετούς εργασίας ε, του πάνελ της ΕΦΣΑ για την ε, διατροφή, για τα διατροφικά προϊόντα και τις αλλεργίες. Υπήρξε υποστήριξη από το προσωπικό της ΕΦΣΑ φυσικά προς το πάνελ και τα μέλη εκτίμησαν ότι περίπου 3.000 προβλήματα που σχετίζονται με τα τρόφιμα από το 2008 μας βοήθησαν χάρη στα στατιστικά δεδομένα να έχουμε πληρέστερα στοιχεία. Με στόχο να προστατεύσουμε τους Ευρωπαίους όσο καταναλωτές ε, να είναι καλύτερα ενημερωμένοι δηλαδή για να κάνουν καλύτερα τις επιλογές τους. Νομίζω ότι χάρη σε αυτές τις προόδους ε, θα, στο μέλλον ε, θα έχω, γίνεται καλύτερα η έρευνα και θα έχουμε περισσότερη καινοτομία. Όπως σας είπα και πέρυσι, μια άλλη βασική συνιστόσα τη εργασίας μας είναι ε, τα πρόσθετα των τροφών με γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί, τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την συσκευασία. Επίσης, είναι σημαντικό να εκτιμήσουμε να αξιολογήσουμε την ασφάλεια, να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα των δράσεών μας καθώς και τις επιπτώσεις επί του ε, περιβάλλοντος. Ε, φυσικά έχουν κυρία σημασία αυτές οι αξιολογίες για την προστασία του κοινού, των καταναλωτών και του περιβάλλοντος, ε, αλλά ταυτόχρονα ε, παρέχουν, προσφέρουν μεγάλη καινοτομία για την εσωτερική αγορά, για την παραγωγή τροφίμων στα πλαίσια της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Αναγνωρίσαμε την ε, σημασία τη πρόοδου που έχουμε σημασία για τα ρυθμισμένα προϊόντα, παραδείγματο χάρη δημιουργία ενό γραφείου αιτήσεων ε, που σε μεγάλο βαθμό θα διευκολύνει τη διάδραση που έχουμε με τους ετούντε και άλλου εμπλεκόμενου φορεί ε, καθώ και την αποτελεσματικότητά μα. Έχουμε φυσικά μειώσει του πόρου που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των βασικών ζητημάτων δημόσια υγεία, αλλά με την αξιολόγηση που κάναμε για αυτά τα ρυθμισμένα προϊόντα καταλήξαμε στο αποτέλεσμα ότι διοχετεύουμε σε αυτό το τομέα περίπου 40% των ετησίων πόρων μας ε, και παρότι ε, έγινε αυτή η αξιολόγηση των τελών για κάποιους τομείς ε, όπου δραστηριοποιείται η ΕΦΣΑ και συνεχίζουμε τον προβληματισμό για αυτό σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά πιστεύουμε ότι για λόγους δημόσιας υγείας θα πρέπει να διατηρηθούν οι πόροι και να ενισχυθούν. τώρα, θα ήθελα να σχολιάσω την, το σχέδιο επιστημονικής στρατηγικής της ΕΦΣΑ για την περίοδο 2012-2016 προς το παρόν είναι αντικείμενο διαβούλευση και τονίζει πόσο σημαντική είναι η προσέγγιση που βασίζεται στην ανάλυση του κινδύνου για την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων ε, του έργου τη ε, ΕΦΣΑ. Εκεί περιγράφονται τέσσερι βασικοί στρατηγικοί στόχοι για το μελλοντικό μα ε, έργο. Θέλουμε να προαγάγουμε έτσι περαιτέρω την επιστημονική μα αριστεία, να βελτιστοποιήσουμε τη χρήση τη ικανότητα αξιολόγηση κινδύνου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να αναπτύξουμε και να εναρμονίσουμε τι μεθοδολογίε αξιολόγηση κινδύνου και να ενισχύσουμε την επιστημονική επιστημονική βάση για την αξιολόγηση κινδύνου και παρακολούθηση αυτού. Εκ παραλλήλου με την επιστημονική στρατηγική έχουμε ε, αναπτύξει μια νέα πολιτική σχετικά με την ανεξαρτησία μεροληψία και επιστημονική ε, διαδικασία λήψης αποφάσεων βασιζόμαστε σε υφιστάμενες ε, προσεγγίσεις, αντλούμε διδάγματα από το παρελθόν και ε, ανεδεικνύουμε σε προτεραιότητα την υψηλή επιστημονική αριστεία. Επίσης, κατέστη δυνατό να κάνουμε μια ευρύτατη διαβούλευση. Επίσης, διοργανώσαμε και ένα εργαστηρίο εδώ στις Βρυξέλλες τον περασμένο μήνα. Ο διάλογος που είχαμε με ένα ευρύτατο κοινό ήταν ιδιαίτερα αξιόλογος και η μεγάλη ποικιλία στις ε, συνεισφορές ε, πιστεύουμε θα εμπλουτίσει την τελική πολιτική και τους εφαρμοστικούς κανόνες. Από αυτή την ε, πλευρά θα ήθελα να ευχαριστήσω την Καρτή Καλιοτάρε που ήταν ο σύνδεσμός μας με τους Ευρωπαίους βουλευτές διότι με την ομιλία τη, ε, έδωσε το ένασμα για την έναξη των εργασιών αυτού του ε, εργαστηρίου. Πριν ε, τελειώσω θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συνεχή υποστήριξη προ το έργο μα και κυρίω ω προ τον προπολογισμό μας. Γνωρίζουμε το δυσχερέστατο οικονομικό πλαίσιο στο οποίο καλείστε εσεί να λάβετε αποφάσει. αλλά πιστεύουμε ότι αν συνεχίσετε να μα υποστηρίζετε θα μπορέσουμε να καλύψουμε τι ανησυχίε και τι προσδοκίε των Ευρωπαίων πολιτών. Είμαι στη διάθεσή σα για οποιοδήποτε ερωτήσεις ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σα ευχαριστούμε πολύ κυρία Διευθύντρια. Ζεστέν Λανέλ. Η υπηρεσία σα ε, πραγματεύεται αυτά τα πολύ σοβαρά θέματα σε ό,τι αφορά την υγεία, την ε, ασφάλεια των τροφίμων, πρόκειται για θέματα που μα αφορούν όλου. Και μετά από το ξέσπασμα του E. coli της περασμένης χρονιάς κατέστησα φες πόσο σημαντικά είναι τα θέματα αυτά. Συζητήσαμε πολύ και θέματα επικοινωνιακής στρατηγικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το πόσα επίπεδα ε, συνακερμού θα πρέπει να υπάρχουν και πώς μπορεί να γίνει καλύτερος συντονισμός. Αναφερθήκατε στα health claims. 3.000, ε. 3.000. Είναι πολύ θετικό το ότι υπάρχουν, ε, υπάρχει διάκριση μεταξύ των επιστημονικά βιώσιμων και μη βιώσιμων τέτοιων αξιώσεων. Και σε ό,τι αφορά θέματα ενημέρωση και ενδεχομένω παραπλάνησης ότι έχει διδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο η ΕΦΣΑ σε ό,τι αφορά την ανεξαρτησία των επιστημόνων των εκτιμητών. Είναι ένα διαρκές θέμα που μας απασχολεί υπήρξε και ένα σχετικό συμπόσιο στις Βρυξέλλες που διοργανώθηκε για να συζητηθεί αυτό το αμφιλεγόμενο θέμα της αξιολόγησης, γιατί φυσικά όλοι μας έχουμε ένα βιογραφικό και όλοι κατά κάποιο τρόπο έχει ασχοληθεί και σε θέματα βιομηχανίας. Αλλά για να απασχολείται κανείς στην Εύσα θα πρέπει να ε, διαπιστωθεί ότι όντω δεν υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα. Τώρα, πολλοί συνάδελφοι έχουν ζητήσει τον λόγο. Θα ήθελα εγώ από πλευρά μου να ρωτήσω θέματα της Βυσσονόλη Α. Το θέμα αυτό έχει καταστεί σημαντικό μετά από την ε, συζήτηση στην ε, Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Θα ήθελα να ρωτήσω πώς έχετε προχωρήσει στην αξιολόγηση της ουσίας αυτής. Η Φρανσουά Γκροστέτ είναι η πρώτη που θα πάρει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μου δίνετε το λόγο. Πάντα χαιρόμαστε πολύ που μπορούμε να έχουμε διάλογο με την Διευθύντρια. Βεβαίω και θα μιλήσω κι εγώ για την διφενόλη Α. Επειδή υπάρχουν διαφορές στην εκτίμηση ανάμεσα στο ευρωπαϊκό επίπεδο και άλλα επίπεδα το γαλλικό για παράδειγμα. Στη Γαλλία, και υπάρχουν πολλά ερωτηματικά βέβαια στην κοινή γνώμη από αυτού, στη Γαλλία λοιπόν έχουμε επιστημονικές γνωμοδοτήσεις και η Γαλλία επιθυμεί να σταματήσει την παραγωγή, την εισαγωγή, την εξαγωγή, τη διάθεση στην αγορά οποιοδήποτε τροφίμου το οποίο περιλαμβάνει διφενόλιο α. Έλεγα λοιπόν ότι ανησυχεί ιδιαίτερα η γνώμη. Γιατί ακούμε ότι η χρήση της ουσίας αυτής μπορεί να είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο ακόμα και όταν ε, προσλαμβάνεται σε πολύ χαμηλές δόσεις. Οι δύο δε εκθέσεις οι οποίες παρουσιάστηκαν στη Γαλλία για την χρήση του χημικού συστατικού αλλά και όσον αφορά την υγεία έλεγε ότι έπρεπε να μειωθεί η έκθεση των πιο ευάλωτων ατόμων, των μικρών παιδιών, των βρεφών ή των γυναικών που θυλάζουν στην ουσία αυτή. Θέλω λοιπόν να ξέρω ποια είναι η δικιά σας η άποψη για τα διάφορα επίπεδα στα οποία καταλήγουν οι εμπειρογνώμονοι. Διαφορετικό στη Γαλλία είπαμε και διαφορετικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα έπρεπε να γίνουν περισσότερες επαφές μεταξύ των διαφόρων αυτών παραγόντων ώστε να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα για τελειώς τα χάνει η γνώμη. Για μένα είναι πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να το ξαναδεί αυτό το θέμα. Δεύτερον, αναφερθήκατε και σε ισχυρισμού όσον αφορά την υγεία. Μας είπατε και εξάλλου έχετε κάνει μια πολύ σημαντική δουλειά επιστημονική, τεράστια και είπατε ότι είναι κάτι που βοηθάει τη βιομηχανία. Θα ήθελα όμως εδώ να δείτε και τον καταναλωτή. Ο καταναλωτής Πού βρίσκεται μέσα σε όλα αυτά. Θα καταλάβει όλες τις πληροφορίες που του δίνετε. Θέλω να ξέρω λοιπόν τη γνώμη σας. Μήπως κινδυνεύουμε να κάνουμε τόσο περίπλοκη την ενημέρωση του καταναλωτή όταν πρόκειται για θέματα που έχουν να κάνουν με τις βιταμίνες ή τα μεταλλικά στοιχεία. Τους ισχυρισμού για την υγεία για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω ότι είναι σημαντικά. Ευχαριστούμε. Λίδα Μακάβεν. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να διευκρινιστεί κάπως το χρονοδιάγραμμα όσον αφορά τους ισχυρισμούς για την υγεία. Θα πάει πριν τα Χριστούγεννα στην Επιτροπολογία. Έτσι είναι. Το 90% των ισχυρισμών αυτών για την υγεία, λένε εφημερίδε, έχουν απορριφθεί από τη βιομηχανία, από τι διάφορε επιχειρήσει. Η σχετική νομοθεσία έχει οθετηθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό για το προφίλ δηλαδή το διατροφικό. Όμως δεν προχωράνε τα πράγματα και ακούγονται, ακούγονται διάφορες διαδόσεις, τι κάνει η Γερμανία στο Συμβούλιο. Είναι αλήθεια αυτά. Δεν μπορούμε να έχουμε, μπορούμε μάλλον να έχουμε μια ξεκάθαρη νομοθεσία και τους συζυγισμούς για την υγεία χωρίς το προφίλ αυτό. Κλούτερ. Ευχαριστώ. Όσον αφορά το διφενόλιο. Δεν πρόκειται μόνο ε, για τα μπιμπερό, πρόκειται και για μεταλλικές κονσέρβες. Επίσης, για τα ζυζανοκτόνια είναι χαμηλότερο τώρα από ό,τι τα πριν από μερικά χρόνια. Καλό αυτό, αλλά υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο συζητάμε. Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα αν συσσωρευτούν. Γιατί εγώ είδα κάποιους ε, ειδικού οι οποίοι είπαν ότι για να αποφύγουμε την υπέρβαση Γι' αυτό χρησιμοποιούνται τώρα διαφορετικά νούμερα για τα ζυζονιοκτόνια. Ποια είναι λοιπόν η λογική αυτή. Προσθέτουμε τελικά τα ποσοστά αν ένα ε, ζυζανοκτόνιο έχει σαν τιμή 40% και ένα άλλο 40% και ένα άλλο 40%. Ε, δεν είναι δυνατόν να τα βάλουμε μαζί γιατί μαζί και τα τρία καταλήγουν στο πάνω από 100%. Η δικιά σας συγγνώμη για την ε, πρόσθεση των τριών αυτών ποσοστών ή όσων είναι τέλο πάντων ποσοστών αυτών, πόσο σα φαίνεται δεν θα καταλήξουμε σε ένα κοκτέιλ ζυζανοκτώνων που θα είναι πολύ πιο επικίνδυνο. Τέτοιε προτάσει σα βρίσκουν σύμφωνοι, τι νομίζετε. Έπειτα. Θυμόσαστε την ανταλλαγή απόψεων που είχαμε στο πάνελ για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Σε τι συμπέρασμα έχετε καταλήξει τώρα. Πώς θα είμαστε σίγουροι ότι θα υπάρχει ενημέρωση όταν το προσωπικό προχωράει. Θα είσαστε περιοριστικοί στην ερμηνεία. Θέλω λοιπόν και γι' αυτά να μου απαντήσετε. Καταλαβαίνετε ότι όπου να είναι θα ληφθούν κάποιες ιδιαίτερα ευαίσθητες αποφάσεις όσον αφορά τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Γι' αυτό και θέλουμε μια καλή αξιολόγηση πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι είναι εντελώ ανεξάρτητοι όλοι οι εμπειρογνώμονε που γνωμοδοτούν όσον αφορά του γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Ευχαριστώ πολύ Κάρλ. Το μέλη αποτελεί εντό ένα θέμα για τον κύριο Πέτερ, που είναι και ο επόμενος που θα πάρει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κοιτάξτε, από τότε που το ΔΕΚ έλαβε μια σαφή απόφαση σε ό,τι αφορά τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς ε, για το μέλι, είμαι σε καλύτερη διάθεση. Θεωρώ ότι τα πράγματα παίρνουν καλύτερο δρόμο. Η ερώτησή μου είναι διαφορετική. Ευχαριστώ ιδιαίτερα την εκτελεστική διευθύντρια για την παρουσίαση αυτή και θεωρώ ότι η υπηρεσία σας συγκαταλέγεται στις πλέον σημαντικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαι όπως πολλοί πολίτες, επεπισμένος ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ του, της ποιότητας των ε, τροφίμων και της υγείας. Και τα πράγματα στην ε, Ευρώπη δυσκολεύουν και παν. Θα ήθελα να μας ε, αναφέρετε τι γίνεται με τους παράγοντες μόλυνσης στην βιομηχανία των τροφίμων. Ποια είναι η επίδραση των λιπαρών ουσιών, των ε, επεξεργασμένων ουσιών στην ε, ποιότητα των τροφίμων. Στην Σλοβενία εντοπίστηκε τρυφίνη σε κάποια έλαια. Και αυτό συνδύεται με τα έλαια των τροφίμων τα οποία είναι επεξεργασμένα. Θα ήθελα να ξέρω κατά πόσο έχετε καταλήξει κάποια συμπεράσματα για το θέμα αυτό και θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχουν και τοποθετήσεις από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ευρωπαϊκή Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ. Ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και την ε, Διευθύντρια και την πολύ ε, ενδιαφέρουσα παρουσίασή της. Χάρηκα ιδιαίτερα γιατί ένα από τα καθήκοντα της ΕΦΣΑ περιλαμβάνει και την προάσπιση των συμφέροντων του Ευρωπαίου πολίτη. Θα ήθελα λοιπόν να αναφερθώ σε κάποια πολύ σημαντικά φαινόμενα και να θέσω και κάποιες ερωτήσεις. Υπάρχει μόλυνση όχι μόνο του εδάφους και του αέρα, αλλά και των τροφίμων και των ζώων εκτροφής στην ε, Βόρεια και στη Βορειοανατολική Ιταλία. Πρόκειται για μόλυνση η οποία προέρχεται από ε, εργοστάσια καύσης και από εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου. Και από τόπους καύσης ε, αποβλήτων. Υπάρχει και ένα εργοστάσιο τσιμέντου στην ε, επαρχία Τρεβίζο της Βενετίας, όπου οι αρωματικοί υδρογονάνθρακες, πολυκυκλικοί υδρογονάνθρακες ε, ήταν διπλάσιοι από το νόμιμο επιτρεπόμενο ποσοστό σε έναν τομέα, σε ένα χώρο, σε μια τοποθεσία που παράγεται το κρασί προσέκο. Και ε, παρουσιάστηκε και ένα σχετικό άρθρο στις εφημερίδες χτες σε ό,τι αφορά δεκαπλάσια ποσά, ποσοστά διοξίνη σε κοτόπουλα από ό,τι επιτρέπεται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Επίσης, στο γάλα της Αγελάδας, σε 18 τοποθεσίες, σε 18 εκτροφές, διαπιστώθηκε μη συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ένα άλλο περιστατικό σε ένα περιφερειακό πάρκο, σε ένα εργοστάσιο τσιμέντου, κοντά σε αγροτικές εκτάσεις. Καταλαβαίνω φυσικά ότι υπάρχουν διαφορετικές, διαφορετικά, διαφορετικές τιμές μόλυνσης σε ό,τι αφορά τα εργοστάσια τσιμέντου. Αλλά σε πολλές περιπτώσεις ε, είναι τριπλάσια, τετραπλάσια, ενιαπλάσια τα ποσοστά αυτά μόλυνσης ε, από σε σχέση μάλλον με, τις, ε, με τους χώρους καύσης αποβλήτων στην Πάρμα. δίπλα στο εργοστάσιο Μπαρίλα υπάρχει τέτοιο εργοστάσιο που για καύση αποβλήτων Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις βιοκαλλιέργειες και την, ε, τους ε, ανησυχούν ιδιαίτερα οι Ευρωπαίοι πολίτες. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν τα σχετικά ε, στοιχεία, γιατί υπάρχουν φυσικά και τα λόμπι των αποτεφρωτών των Δήμων και Κοινοτήτων που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Θα πρέπει λοιπόν να γίνουν σωστές αναλύσεις και τα αποτελέσματα είναι πραγματικά αρνητικά και σε ό,τι αφορά τα κοτόπουλα με διοξίνη. Τα πράγματα ήταν πολύ ανησυχητικά. Να ρωτήσω λοιπόν την Διευθύντρια κατά πόσον η ΕΕΦΣΑ δεν θα μπορούσε να εξετάσει στα σοβαρά να διεξάγει μια μελέτη για τι επιπτώσεις ε, των αποτεφρωτήρων και των εργοστασίων τσιμέντου στις ε, γεωργικέ καλλιέργειες και στις εκτροφέ ζώων προκειμένου να προστατεύσει τα συμφέροντα των πολιτών και των καταναλωτών. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε πραγματικά να δώσουμε απαντήσεις στα μεγάλα ερωτηματικά που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στις περιφέρειες αυτές. Uh, Κρήτον είναι uh, Καλώς ήρθατε. Πολλά θέματα ετέθησαν ήδη όσον αφορά την ανεξαρτησία της ΕΦΣΑ. Συχνά στην αίθουσα αυτή καθόμαστε και συζητάμε για... ή παίρνουμε αποφάσεις που δεν είχαμε λόγο να πάρουμε αν ξέραμε ότι η ΕΦΣΑ είχε μια πραγματική ανεξαρτησία και μπορούσε εντελώ ανεξάρτητα να φέρει σε πέρα στα καθήκοντά της. Ίσχυε και για άλλα θεσμικά όργανα. για οργανισμούς που κάνουν αξιολογήσεις και το έχουν πει πολλοί. Ενημερώνεται η ΕΜΑ, για παράδειγμα, από κάποιον ότι υπάρχει μια διαφωνία. Και τι κάνουνε, αλλάζουνε το άτομο αυτό. Ότι εμείς όμως θέλουμε αντίθετα να στηρίζουν τα άτομα αυτά. Όχι να κρύβονται πράγματα. Θα ήθελα λοιπόν να σχολιάσετε ακριβώς αυτό. Καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί στρεβλώσεις όσον αφορά την πολιτική μας δουλειά. Αν έχουμε έναν οργανισμό ο οποίος συνεχίζει να δημιουργεί αμφιβολίες όσον αφορά την ανεξαρτησία του. Μα είναι τόσο δύσκολο τελικά να απομακρύνεται άτομα από τις επιτροπής, από την εκάστοτε επιτροπή, άπαξ και υπάρχει απόδειξη ε, ότι, είναι, ότι μπλέκονται συμφέροντα, ότι υπάρχει το ασυμβίβαστο. Θα ακούσουμε τις απαντήσεις, λέει ο Πρόεδρος. Ωστόσο, και εγώ κάποιες φορές έχω την εντύπωση ότι υπάρχει μια στρατηγική για ίδιους σκοπούς. Ε, διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν προβλήματα στην ΕΦΣΑ και τα προβλήματα αυτά συνεχίζουν παρά το γεγονός ότι άλλαξε η πολιτική. Έχουμε εδώ και τηλεοπτικές, ε, τηλεοπτικά κανάλια που θέλουν να ακούσουν πώς θα διασφαλίσουμε και πώς εκτιμούμε την ανεξαρτησία της ΕΦΣΑ. Θα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι ε, έχει υπάρξουν, αλλά, ότι έχουν υπάρξει αλλαγέ και να μην ε, επανελχόμαστε σε προβλήματα που υπήρχαν πριν από χρόνια. Θα ακούσουμε όμω τι απαντήσει σα. Ο κύριο Ζέμπερ. Ναι, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω, Γιώ, για αυτή τη διευκρίνηση, γιατί και εγώ το ίδιο πιστεύω. Υπήρχαν προβλήματα, αλλά νομίζω ότι για θέματα ανεξαρτησία θα πρέπει να είναι σαφέ. Μόνο όταν κάποιο έχει δουλέψει για κάποιο χρονικό, μα, μάλλον το γεγονό ότι κάποιο έχει δουλέψει για κάποιο χρονικό διάστημα για κάποιο όμιλο, δεν σημαίνει ότι δεν είναι ανεξάρτητο. Γιατί, για παράδειγμα, όταν κάποιο έχει δουλέψει για μία μη κυβερνητική οργάνωση, δεν σημαίνει αυτό ότι για πάντα μετά είναι άχρηστο για κάποιου σκοπού. Όχι, θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια. Θα πρέπει να υπάρχουν εγγύησει από το εκάστοτε άτομο ότι πρόκειται να εκτελέσει τα καθήκοντά του με ανεξαρτησία. Το να αποκλείσουμε ένα άτομο για την θεωρούμε ότι δεν είναι ανεξάρτητο επειδή κάποτε είχε εργαστεί, θεωρώ ότι είναι μη ρεαλιστικό. Σας το λέω ξεκάθαρα. Θεωρώ ότι οι υπηρεσίες όπως η ΕΦΣΑ προσλαμβάνουν άτομα τα οποία απασχολούνται στον εκάστοτε τομέα και αυτό περιλαμβάνει και την βιομηχανία και θεωρώ ότι είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε ότι θα εκτελούν τα καθήκοντά τους με ανεξαρτησία και εδώ θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχουν εγγύησει. Αλλά τώρα να καταδικάσουμε κάποιον ε, στην αιωνιότητα θεωρώ ότι είναι μη ρεαλιστικό. Γιατί δεν ανταποκρίνεται και στις επιθυμίες μας στην τελική ανάλυση. Μία δεύτερη ερώτηση προς την κυρία Διευθύντρια. Ποια είναι τα βασικά διδάγματα από το ξέσπασμα της κρίσης η κόλαη. Εγώ θεωρώ ότι έφταγε η διαχείριση της πληροφορίας, των πληροφοριών για τις ζημιές που υποστήκαμε και νομίζω ότι θα έπρεπε η ΕΦΣΑ να εξαγάγει συμπεράσματα για το πώς μπορούν να συντονιστούν οι εθνικές πολιτικές προκειμένου να μην δημιουργείται τέτοια εξαιρετική ανασφάλεια στους ε, καταναλωτές. Υπήρξε, όπως σας ανέφερα, εξαιρετική πολλές ζήμιες χωρίς αυτό να διασφαλίσει την ασφάλεια του καταναλωτή και αυτό θεωρώ ότι μπορούμε να το βελτιώσουμε κάτι άλλο σε ό,τι αφορά τους γενετικά τραποποιημένους οργανισμούς όπως είπε και ο Κάρλ Σλούτερ. Ακούω διαρκώς ότι η ΕΦΣΑ δεν ελέγχει όλο το φάσμα των κινδύνων σε ό,τι αφορά τον περιφερειακό χαρακτήρα των κινδύνων σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπο στο φυσικό περιβάλλον σε, κάποια, σε κάποιους χώρους. Τι μπορείτε λοιπόν να πείτε για αυτό το θέμα, για το εύρος του φάσματος των ε, μελετών της ΕΦΣΑ, ότι καλύπτει όλη την Ένωση και ότι δεν περιορίζεται χρονικά τοπικά. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν σημαντικό να το γνωρίζουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η Σοφή Οκουνή. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κυρία Διευθύντρια, χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχουμε εδώ. Αλλά λυπάμαι πραγματικά που δεν είμαστε πιο πολυάριθμοι για να έχουμε μια πραγματική συζήτηση εδώ μαζί σας. Τώρα διάφορα θέματα ετέθησαν και έχω να σας μεταφέρω ορισμένες σκέψεις για το διφενόλιο α πρώτα απ' όλα. Όσον αφορά την ουσία αυτή, ο βαθμός επικινδυνότητας και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται επικίνδυνη η ουσία αυτή είναι κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε ακόμα αρκετά καλά. Καταλαβαίνουμε βέβαια ότι μεταλλάσσεται στα τρόφιμα όταν θερμαίνονται τα υλικά ε, στα οποία περιλαμβάνονται τα τρόφιμα σε ένα πλαστικό δηλαδή το οποίο το βάζουμε στο φούρνο μικροκυμώτων, τότε η διφενόλη περνάει στα τρόφιμα. Δεν είναι λοιπόν δικό σας ρόλος, και είναι πραγματική ερώτησή μου αυτή, δεν είναι δικό σας ρόλος να ζητήσετε αυτή η κατάσταση, αυτό το φαινόμενο να αναφέρεται στις συσκευασίες Δηλαδή να λέμε ξεκάθαρα στον καταναλωτή ότι κοιτάξτε το προϊόν αυτό που αγοράζετε, αν το θερμάνετε πρέπει να το ζεστάνετε σε ένα γυάλινο δοχείο και όχι σε ένα πλαστικό. Αυτό ήταν το πρώτο για το διφενόλιο. Δεύτερον, ε, μετά το παραμπαίνει στα καλλιντικά, η ασπαρτάμι, είναι ένα προϊόν το οποίο επίσης τίθεται υπό φυσβήτησε όλο και περισσότερο τον τελευταίο καιρό ως καρκινογόνο. Ο οργανισμός σας δουλεύει πάνω σε αυτό. Εγώ σε αυτή την επιτροπή έχω έρθει πρόσφατα σχετικά και δεν ξέρω. Έχετε ήδη ξεκινήσει εργασίες σχετικά με το προϊόν αυτό. Υπάρχουν ε, κάποια σχέδια, έχετε κάποιες σκέψεις πάνω σε αυτό. Τέλος, διοξίνες. Οι δύο διοξίνες, ορισμένα προϊόντα προς κατανάλωση, που προέρχονται από τη Σουηδία, αν δεν απατώμε, και που εξάγονται στις διάφορες χώρες μέλη, χωρίς όμως να αναφέρεται στα προϊόντα αυτά ε, ρητά ότι το ποσοστό διοξίνης είναι ιδιαίτερα υψηλό, το οποίο περιέχεται στα προϊόντα αυτά. Δεν θα έπρεπε να γνωρίζει ο καταναλωτής καλύτερα τι καταναλώνει, ακόμα και αν τα προϊόντα αυτά έχουν τιμές διοξίνης υψηλά, γιατί βλέπετε εξαρτάται από το τι ήθιστε στις χώρες από τις οποίες εξάγονται αυτά τα προϊόντα και εκεί μπορεί να είναι ανεκτό ένα υψηλότερο ποσοστό περιεκτικότητας διοξινών. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Πολλές οι ερωτήσεις σας. Θα ξεκινήσω με το διφενόλιο. Μια που με ρωτήσατε πολύ πάνω σε αυτό. Εδώ έχω να σας πω λοιπόν το εξής. Αναγνωρίζω πρώτα απ' όλα ότι είναι ένα ιδιαίτερα επίμαχο θέμα και πολύ σωστά αναφέρατε ότι πρόσφατα έχουν γίνει δημοσιεύσεις από την Γαλλική Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας Τροφίμων πάνω σε αυτό. Κατά το παρελθόν είχαμε και άλλες τέτοιες δημοσιεύσεις. Δεν είναι δηλαδή η πρώτη φορά που βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια τέτοια διαφωνία ε, μεταξύ διαφόρων εθνικών αρχών πάνω στο προϊόν αυτό. Γι' αυτό εξάλλου και ε, ο Παγκόσμιο Οργανισμός Υγείας πέρυσι οργάνωσε ένα εργαστήριο στο οποίο συμμετείχαν πολλές χώρες με εκπροσώπου και από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων ακριβώς με αυτό το αντικείμενο. Και θα θυμόσαστε ότι δημοσίευσαν ε, στα τέλη τη προηγούμενης χρονιάς την έκθεσή τους, συγγνώμη διορθώνω μιλήτρα την Άνοιξη φέτο. Και το συμπέρασμα ευθυγραμμίζεται με τα συμπεράσματα του πάνελ της ΕΦΣΑ. Τώρα για να έρθω πάλι στις ε, εκθέσεις της γαλλικής υπηρεσίας για παράδειγμα. Εμείς δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Πιστεύουμε ότι για μας είναι πάντα σημαντικό όταν έχουμε νέα επιστημονικά δεδομένα να αναθεωρούμε ε, τα συμπεράσματά μας, να δούμε κατά πόσο δηλαδή τα νέα αυτά δεδομένα ε, πρέπει να αλλάξουν τα δικά μας συμπεράσματα. Το ίδιο ισχύει λοιπόν και με αυτή την έκθεση. Θα καταλήξουμε για το κατά πόσο πρέπει να αλλάξουμε ή όχι την δικιά μας ε, γνωμοδότηση, την οποία δημοσιεύσαμε πριν από ένα χρόνο, που ήταν μια αξιολόγηση κινδύνου όσον αφορά το διφενόλιο. Τώρα, ε, για μένα είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή να σας πω ε, ποια είναι τα συμπεράσματά μας, μια που είχαμε τη δημοσίευση τέλη Σεπτεμβρίου. Το πάνελ μας δουλεύει πάνω σε αυτήν. Όμως επιτρέψτε μου να αναφέρω ότι οι δύο εκθέσεις δεν είναι αυτό που θα ονομάζαμε εμείς αξιολόγηση κινδύνου. Υπάρχει μία, όπως είπατε κι εσείς, η οποία περιγράφει την έκθεση στο διφενήλιο ε, από τον γαλλικό πληθυσμό και η άλλη ε, συμπεριλαμβάνει πιο πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα για τη διφενήλιο. Το πάνελ μας λοιπόν θα δουλέψει πάνω σε αυτά. Σε συνεργασία μάλιστα με Γάλλους ειδικού. Έχουμε ξεκινήσει δηλαδή διάλογο. Καταλαβαίνουμε τι λέει η έκθεση, ε, τα συζητάμε μαζί τους, δεν καθόμαστε απλώς να διαβάσουμε την έκθεση, κάνουμε συζήτηση μαζί τους. Και στόχος μας είναι να ετοιμάσουμε και να δημοσιεύσουμε τελικά μια κοινή, από κοινού έκθεση με τις γαλλικές αρχές, όπου θα εξηγούμε που συμφωνούμε και που όχι και γιατί. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό για να μην υπάρχουν αυτές οι διαφωνίε, όπως είπατε. Αυτό θα γίνει τέλη Νοεμβρίου. Θα δημοσιεύσουμε την ε, ε, κοινή αυτή έκθεση και θα κάνουμε και μια επιστημονική δήλωση που θα βασίζεται στην έκθεση αλλά και στα τελευταία επιστημονικά δεδομένα που θα έχουμε για το διφενήλιο. Γιατί κάθε μέρα έχουμε καινούρια. Έχουμε 10 τουλάχιστον νέες επιστημονικές δημοσίευσεις. Οπότε ποτέ δεν ξέρουμε. Σύντομα λοιπόν, σας ενημερώνω ότι παίρνουμε πολύ σοβαρά την έκθεση αυτή. Μιλάμε με τους Γάλλους εμπειρογνώμονες και θα σας ενημερώσουμε για το αποτέλεσμα των εργασιών μας σε μερικές εβδομάδες από τώρα. Και επειδή αναφέρομαι στο Δεφινέλιο, θέλω επίσης να σας πω ότι βάση για την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για προϊόντα που χρησιμοποιούνται στις συσκευασίες, Εάν κάποια συστατικά από τη συσκευασία περνάνε στα τρόφιμα, η ουσία που μεταφέρεται δεν θα πρέπει να οδηγεί σε κανένα πρόβλημα για την υγεία. Δεν λέω ότι ισχύει για το συγκεκριμένο συστατικό, αλλά μερικές φορές έχετε συστάσεις επιπλέον. Έχετε δηλαδή σε ορισμένες συσκευασίε συστάσεις για το πώς πρέπει να χρησιμοποιείτε ή τι πρέπει να αποφύγετε στην χρήση ε, του τροφίμου αυτού. Τέτοιες συστάσεις δηλαδή γίνονται πολλές φορές προς τον πληθυσμό. Ε, τώρα ισχυρισμοί για την υγεία. Ελπίζω ο καταναλωτής να καταλήξει, γιατί η επιστημονική δουλειά που έχουμε κάνει μέχρι τώρα έχει ως στόχο την καλύτερη προστασία των καταναλωτών και ιδιαίτερα ε, θέλει να τους βοηθήσει να κάνουν καλύτερες διατροφικές επιλογές. Πρέπει να σας πω ότι σήμερα στην αγορά είναι τόσο πολλοί ισχυρισμοί σχετικοί με την υγεία που φυσικά και είναι δύσκολο. Μετά τη δουλειά της ΕΦΣΑ πάντως γιατί 80% των ισχυρισμών υγείας ε, που έχουμε αξιολογήσει έχουν απορριφθεί. Αλλά θα τελειώσουμε εφόσον η Επιτροπή, όπως είπε και η Λίντα Μακάβιν, εφόσον η Επιτροπή έχει καταλήξει με τα κράτη-μέλη σε ένα θετικό κατάλογο ισχυρισμών για την υγεία. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι αυτό θα γίνει στα τέλη της χρονιάς τότε θα έχουμε τη σχετική πρόταση. Θα είναι πολύ σημαντικός αυτός ο κατάλογος. Επίσης θέλω να αναφέρω ότι στην ΕΦΣΑ ακόμα πρέπει να αξιολογήσουμε διάφορα βότανα, κάπου 1500 σχετικά με τα οποία υπάρχουν επίσης ισχυρισμοί για την υγεία. Και περιμένουμε γιατί η Κομισιόν είπε ότι χρειάζεται χρόνο για να σκεφτεί πάνω σε αυτά, διότι ίσως υπάρξει μια δυσκολία στην εφαρμογή των κανόνων. Θεωρεί ότι τα προϊόντα αυτά μπορεί να έχουν χρήση είτε στην ιατρική, είτε να είναι βότανα, τα οποία χρησιμοποιούνται στη μαγειρική. Οπότε πρέπει να δούμε τι ευρωπαϊκή νομοθεσία προβλέπεται και να μην υπάρξει παρεξήγηση ή σύγχυση για τους καταναλωτές με τα βότανα. Οπότε περιμένουμε ακόμα, εκκρεμεί αυτή η υπόθεση δηλαδή. Τώρα για το διατροφικό προφίλ. Ζητήσαμε επιστημονική γνωμοδότηση πριν από λίγο καιρό. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε σύντομα εφόσον έρθει η Επιτροπή με κανόνες για την εφαρμογή του προφίλ αυτού, αυτό λοιπόν που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι να δούμε κατά πόσο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάτι σαν ένα καλάθι τέτοιων προϊόντων και τέτοιων προφίλ και ίσως έτσι μπορέσουμε να βοηθήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να ξεκινήσει μια αξιολόγηση του διατροφικού αυτού προφίλ σχετικά με την σήμανση και τους ισχυρισμού για την υγεία των προϊόντων. Ζήσανε οκτώνια τώρα. Αυτό που λέτε είναι ορθά, ότι δηλαδή όταν ιδιαίτερα στην έκθεση στην οποία αναφέρθηκα πριν λέμε ότι υπάρχει παρουσία υπολείπων και ποιο είναι το ανώτατο επίπεδο υπολείπων Αυτό ισχύει για όλα τα ζυζανιοκτόνια. Ξέρουμε ότι για τους καταναλωτές αυτό σημαίνει ότι μπορεί να είναι διαφορετικές ουσίες και όχι μόνο μία ε, που αφήνει υπόλοιπα ε, στην τροφή τους. Αυτό λοιπόν πάνω στο οποίο δουλεύουμε στην ΕΦΣΑ είναι το εξή. Θέλουμε να προχωρήσουμε περισσότερο όσον αφορά την μεθοδολογία, να αναπτύξουμε περισσότερο την ε, μεθοδολογία μας, ιδιαίτερα για την συσσωρευτική αξιολόγηση, που σημαίνει ότι δεν κοιτάμε μόνο μία ουσία και τις επιπτώσεις της στην υγεία, αλλά και τον συνδυασμό που μπορεί να επηρεάζει η... μία ουσία την επιρροή της άλλης ή να την εξωτερώνει σε έναν βαθμό. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε μια επιστημονική γνωμοδότηση πάνω σε αυτό. Πιστεύουμε λοιπόν ότι στα τέλη του 2012 θα είμαστε σε θέση να χρησιμοποιήσουμε την μεθοδολογία αυτή για τα συσσωρευτικά υπόλοιπα σε καθημερινή βάση. Είναι ένα δύσκολο επιστημονικά θέμα, έχουμε όμως επενδύσει πολύ. Έχουμε συνεργαστεί και με άλλους εταίρους σε διεθνές επίπεδο και θα χρησιμοποιήσουμε ε, τη μεθοδολογία αυτή, ελπίζω από του χρόνου, στην ε, καθημερινή μας ρουτίνα αξιολόγηση. Έρχομαι τώρα στο θέμα της ανεξαρτησίας. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ όλους εσάς που σε συνεχή βάση δουλεύετε πάνω σε αυτά τα θέματα και βοηθάτε να έχουμε πρόοδο. Τι θέλω να πω είναι ότι η πολιτική μας κάθε φορά που υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων εδώ και δέκα χρόνια είναι ότι παρόλο που ενισχύθηκαμε το 2007 μπορώ να πω ότι έχουμε μια καλή εμπειρία και ότι κάθε χρόνο τουλάχιστον σε τρεις περιπτώσεις αποκλείουμε πλήρως ή μερικώς εμπειρογνώμονες από τις δραστηριότητές μας. Όταν ανανεώνουμε τα πάνελ μας, όταν επιλέγουμε εμπειρογνώμονες για ομάδες εργασίας, ε, φυσικά και ελέγχουμε ώστε να μην υπάρξει ενδυνάμει σύγκρουση συμφερόντων. Και κάνουμε και screening 5.000 δηλώσεις συμφερόντων το χρόνο. Πρέπει όμως να αναγνωρίσουμε ότι παρόλο που έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια και παρόλο που έχουμε δουλέψει πολύ σκληρά πάνω σε αυτό, πρέπει να συνεχίζουμε να αναθεωρούμε την πολιτική μας. Και αυτό που κάνουμε με τη νέα πολιτική μας που συζητήσαμε τον Οκτώβριο στο εργαστήριο αυτό που οργανώσαμε εδώ στις Βρυξέλλες είναι ότι πρέπει και να μάθουμε από τις εμπειρίες μας αλλά και να καταλάβουμε ότι το θέμα της ανεξαρτησίας δεν είναι μόνο η διαχείριση της σύγκρουσης συμφερόντων. Σίγουρα αυτό αποτελεί ένα σημαντικό πυλώνα για να έχουμε ανεξαρτησία. Πιστεύουμε όμως ότι υπάρχουν και άλλοι πυλώνες με ποιο τρόπο επιλέγουμε τους εμπειρογνώμονες, για παράδειγμα. Με ποιο τρόπο συλλογικά λαμβάνονται οι αποφάσεις συμπεριλαμβανομένων όλων των μελών των πάνελ ή των ομάδων εργασίας. Δεν πρόκειται δηλαδή για την γνωμοδότηση ενός εμπειρογνώμονος ποτέ. Είναι συλλογικό έργο που απορρέει από μια συλλογική, από μια συζήτηση, μια συλλογική διαδικασία. Φυσικά και γίνεται screening των συμφερόντων εσείς μπορεί να δείτε ότι κάποιος δυνάμει μπορεί να οδηγηθεί σε σύγκρουση ε, συμφερόντων, το άτομο αυτό δεν πρόκειται ποτέ να υπογράψει από μόνο του την όποια γνωμοδότηση. Η γνωμοδότηση απορρέει από μια συλλογική διαδικασία. Φυσικά και έχουμε πολιτική για την ανεξαρτησία και αυτή είναι το ότι ξεκαθαρίζουμε σε όλους ότι οποιοδήποτε τροποποιεί επιστημονικά ε, δεδομένα, φυσικά και είναι κάτι που προσέχουμε να μην απορρέει από σύγκρουση συμφερόντων, αλλά ότι έτσι κι αλλιώς υπάρχει διαφάνεια και υπάρχει και συλλογική δουλειά. Ο τρόπος με τον οποίο συλλέγονται επίση τα δεδομένα είναι τέτοιος που δεν μπορεί να υπάρξει στρέβλωση. Όλα αυτά λοιπόν τα κάνουμε με την νέα μας πολιτική. Θέλουμε βέβαια να κάνουμε ακόμα περισσότερα, γιατί αναγνωρίζουμε ότι αντιμετωπίζουμε μια πρόκληση όσον αφορά την ανεξαρτησία μας. Στο εργαστήριο αυτό λοιπόν που οργανώσαμε τον Οκτώβριο, από αυτή την άποψη πρέπει να πω ότι είχαμε πολύ ε, ενδιαφέρουσες συζητήσεις και συμπεράσματα. Αποτελεί πια έναν ακρογωνίο λίθο για μας όσον αφορά την οργάνωσή μας, τη σχέση μας με τη βιομηχανία, πόσο επιλέγουμε τους επιστήμονες, τους εμπειρογνώμονες από τα κράτη-μέλη. Ξέρουμε ότι η ανεξαρτησία έχει να κάνει και με το πώς την αντιλαμβάνεται κανείς. Το αποτέλεσμα λοιπόν του εργαστηρίου αυτού και η δημόσια διαβούλευση που ξεκινήσαμε τον προηγούμενο μήνα θα μας οδηγήσει στο να λάβουμε υπόψη μας νέα σχόλια στην πολιτική μας και να εφαρμόσουμε νέους κανόνες. Πράγμα το οποίο θα υποβάλουμε το Δεκέμβριο στο ε, Διοικητικό μας Συμβούλιο. Τώρα, για το άλλο πολύ σημαντικό θέμα που αναφέρεται και που έχει να κάνει με το προσωπικό. Έχουμε ειδικού κανόνες έτσι ώστε να διασφαλίσουμε όχι μόνο ότι οι εξωτερικοί πυρογνώμονες ε, δεν θα διηγηθούν σε σύγκρουση συμφερόντων, αλλά ο ίδιος κανόνες ισχύει και για το προσωπικό μας, όταν προσλαμβάνονται, όταν δουλεύουν στην ΕΦΣΑ και όταν φεύγουν από την ΕΦΣΑ επίσης. Υπάρχει ο κανονισμός προσωπικού, ο οποίος διέπει όλους μας. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο είναι ότι ζητάμε από το εκτελεστικό μας προσωπικό κάθε χρόνο να υπογράφει μία δήλωση συμφερόντων. Να την ενημερώνει κάθε χρόνο. Η οποία ελέγχεται από τους ε, ανώτερους έτσι ακριβώς ώστε να μην υπάρχει τέτοια σύγκρουση συμφερόντων. μετά από κάποια χρόνια ορισμένοι φεύγουν από την ΕΦΣΑ και ανανεώνονται ή δεν ανανεώνονται κάποια συμβόλαια. Οπότε τώρα έχουμε πιο δυνατέ διαδικασίες, ώστε όταν φεύγει κάποιος από την ΕΦΣΑ, να μην φεύγει για να πάει σε έναν οργανισμό ο οποίος εν δυνάμει θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει πληροφορίες που διαθέτουν οι υπάλληλοι μας. Να μην υπονομεθεί το απόρριτο από την ΕΦΣΑ και καταλήξει στη βιομηχανία. Έχω ένα παράδειγμα πολύ πρακτικό. Πριν από λίγο καιρό έφυγαν ορισμένοι από την ΕΦΣΑ και πήγαν στη βιομηχανία. Εμείς βάλαμε προϋποθέσεις να μην υπάρχει σχέση με το προσωπικό μας, με τους εμπειρογνώμονες ε, πια, έτσι ώστε να μην μπορεί εν δυνάμει να υπάρξει σύγκρουση συμφερόντων ανάμεσα στις δραστηριότητές τους που είχαν στην ΕΦΣΑ και τις δραστηριότητές τους σε άλλες Οπότε, το στοιχείο κλειδί εδώ είναι ότι καθημερινά ασχολούμαστε με αυτό και τακτικά να θεωρούμε την πολιτική μας και η νέα μας πολιτική θα βασιστεί στους υπάρχοντες κανόνες και στην εμπειρία που έχουμε συλλέξει κατά το παρελθόν. Τι μαθήματα πήραμε από το e-coli, από την κρίση αυτή πολλά μαθήματα. Πρώτα απ' όλα, έδειξε, όπως είπα και νωρίτερα, ότι σωστά ετοιμάζουμε την υπηρεσία μας για τέτοιου είδους κρίσεις. Και εδώ δεν μιλάω μόνο για τις διαδικασίες, αλλά για τα δίκτυα που έχουμε τις εθνικές υπηρεσίες ασφαλείας τροφίμων, με διεθνείς οργανισμούς, ε, το ότι συλλέγουμε στοιχεία, γιατί δεν είναι κατά τη διάρκεια μιας κρίσης που θα συλλέξουμε στοιχεία, πρέπει από πριν να τα έχουμε συλλέξει. Και μπορούμε επίσης να δοκιμάσουμε έτσι και τη δυνατότητά μας ε, αντιμετώπισης μιας κρίσης, κάτι το οποίο κάνουμε κάθε χρόνο με την Επιτροπή. Τι άλλο μάθαμε. Ότι πρέπει να συνεχίσουμε να επενδύουμε ε, στα θέματα του κατεπήγοντος. Δεν είναι ότι δεν ξέραμε για το e-coli. Δυστυχώς η Ευρώπη είχε εμπειρία με ξεσπάσματα τέτοιων κρίσεων και παλιότερα. Τι δείχνει όμως. Δείχνει ότι είναι σημαντικό και εδώ είναι που η ΕΦΣΑ μπορεί να προσφέρει μια προστιθέμενη αξία στο σύστημα ότι πρέπει να συνεχίσουμε να ενημερώνουμε καλύτερα τη βάση δεδομένων μας και με τα δίκτυα που έχουμε στις 27 χώρες, προκειμένου να προλαμβάνουμε εν δυνάμει προβλήματα σαν κι αυτό. Μάθαμε επίσης ότι η παραγωγή σπόρων επίσης και βλαστών είναι κάτι ε, το οποίο λοχεύει κινδύνους και ότι πρέπει να το διαχειριστούμε καλύτερα στο μέλλον. Γι' αυτό και δουλεύουμε πάνω σε μια αξιολόγηση κινδύνου πάνω στα προϊόντα αυτά για να μπορούμε να δώσουμε τη γνωμοδότησή μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία στη συνέχεια να καθορίσει κανόνες ώστε να αποφεύγονται τέτοιες καταστάσεις στο μέλλον. Γιατί την Πράγματι, ναι, δουλεύουμε πάνω στην ασπαρτάμε. Η Ασπαρτάμι ήταν στο πρόγραμμα εργασίας μας, αλλά επειδή υπήρξαν πάρα πολλές ανησυχίες, ήταν για το 2018, πολύ αργότερα, αλλά επειδή είχαμε κάποια στοιχεία, η Επιτροπή μας ζήτησε να κάνουμε την αξιολόγηση κινδύνου για την ασπαρτάμι πιο νωρίς. Γι' αυτό και θα κάνουμε μια πλήρη αξιολόγηση κινδύνου όσον αφορά την ασπαρτάμι, που θα είναι έτοιμη στα τέλη της επόμενης χρονιάς, πιστεύω. Ξεκινήσαμε με μια συλλογή δεδομένων. Ε, πήραμε επιστημονικές μελέτες και δημοσιευμένα στοιχεία και πρόκειται να δημοσιεύσουμε τα δεδομένα αυτά όταν θα ξέρουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι είναι αυτό εφικτό. Θα δημοσιεύσουμε όλα τα στοιχεία τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε για να καταλήξουμε στην αξιολόγηση κινδύνου για την Ασπαρτάμι. Θα είναι δηλαδή στη διάθεση του κοινού το Δεκέμβριο. Στη συνέχεια κάνουμε μια ομάδα εργασίας από το πάνελ μας για τις πρόσθετες ουσίες. Θα φροντίσουμε να προσφέρουμε στοιχεία και δεδομένα τα οποία θα κάνουν το κοινό να εμπιστεύεται ακόμα περισσότερο τα προϊόντα που καταναλώνει. Σκοπεύουμε να έχουμε και μια δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο έκθεσης που θα έχουμε ετοιμάσει για την Ασπαρτάμι του χρόνου. Την άνοιξη κατά πάσα πιθανότητα στις αρχές του καλοκαιριού. Ώστε για ένα τόσο επίμαχο επιστημονικά θέμα να έχουμε όσο γίνεται περισσότερα στοιχεία. Γι' αυτό και θα ζητήσουμε από την Κομισιόν να καθυστερήσει λίγο ε, την δημοσίευση ώστε να προλάβουμε να έχουμε μια εκτενή διαβούλευση. Δύο ξύνες τώρα, αυτό είναι το τελευταίο μου. Ελπίζοντα ότι δεν θα ξεχάσω. Α, είπατε να και για το ΜΕΛΗ και για του γενικά του οργανισμούς. Λοιπόν, για τι δύο Πρώτα απ' όλα πρέπει να σας πω, επειδή πολλοί με ρωτήσατε, εξαιτία της ε, μόλυνσης, της επιμόλυνσης και των διοξινών και των ε, PCB, των πολυχλωριωμένων διφενηλίων, υπάρχουν, υπάρχει, μάλλον υπάρχουν μέτρα ε, όσον αφορά τις διοξίνες. Το ξέρουμε αυτό. Ξέρουμε ότι είναι καρκινογενείς οξύνες, γι' αυτό και πρέπει να προλαμβάνονται ε, περιπτώσεις κατανάλωσης τροφίμων που περιέχουν παραπάνω από τα ανώτατα επιτρεπτά ε, ποσά, ποσοστά. Πρέπει να αφαιρούνται από την αγορά τέτοιου είδους τρόφιμα. Χρησιμοποιούμε πάντως τα στοιχεία τα οποία συλλέγουν τα κράτη-μέλη, τα 27. Συλλέγουμε όλα τα δεδομένα, διότι έχουμε ένα πρόγραμμα εποπτείας στα κράτη-μέλη και κάθε χρόνο ετοιμάζουμε έκθεση για το επίπεδο επιμόλυνσης των τροφίμων και των ζωοτροφών με διοξίνες. Είναι μια πολύ σημαντική δουλειά αυτή. Βοηθάει να ε, γνωρίζουμε και καλύτερα πού βρισκόμαστε όσον αφορά την μείωση της παρουσίας ε, διοξίνης αυτού του, αυτής της ουσίας που τόσο παρουσιας διοξινης αυτου του αυτης μολύνει τα τρόφιμά μας. Η κατάσταση πάντως πρέπει να ξέρετε ότι σήμερα είναι καλύτερα από ό,τι ήταν πριν από 15 χρόνια εξαιτίας των δράσεων που έχουν αναλυφθεί μέχρι τώρα. Πρώτα απ' όλα η απαγόρευση ορισμένων χημικών ουσιών στη βιομηχανία γενικά, όχι μόνο τρόφιμα, στη βιομηχανία γενικά, αλλά και επειδή ελέγχουμε και υπάρχει και ευρωπαϊκή νομοθεσία ιδιαίτερα αυστηρή όσον αφορά τα ανώτατα επίπεδα παρουσίας διοξινών. Αυτά λοιπόν είναι θέματα τα οποία τακτικά δημοσιεύουμε και έτσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να βρει Όσον αφορά τώρα το μέλι, μαζί ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, όπως είπατε και εσείς, να πούμε κατά πόσο πιστεύουμε ότι το μέλι που περιλαμβάνει γύρι το μόνο α10 από το συμβατικό καλαμπόκι. Μέσα στο λίγο χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μας μπορέσαμε να βρούμε στα στοιχεία που δόθηκαν όχι ότι είναι ασφαλής μεν, αλλά ότι δεν υπάρχει επιπλέον κίνδυνος ανάμεσα στην γύρι από το συμβατικό καλαμπόκι και την γύρι από το μόν α10. Εννοείται ότι στο μέλλον, αλλά δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα το αποφασίσουμε, περιμένουμε ότι θα συζητηθούν και άλλα στοιχεία όσον αφορά την ε, παρουσία ε, της γύρης. Θα πρέπει ασφαλώς να αξιολογήσουμε πολύ περισσότερο το θέμα των επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία από την γύρη. Δεν ξέρω αν ξέχασα κάτι, αλλιώς ευχαρίστως να επανέλθω. Ναι, υπάρχει, θα εργοπορήσουμε γιατί πρέπει να περιμένουμε μέχρι τις 5 όπως λέγαμε, οπότε γιατί να κάνουμε διάλειμμα και να μην κάνουμε ένα δεύτερο γύρο ερωτήσεων αν θέλετε, παρακαλώ. Eh, Ευχαριστώ. Άκουσα την απάντησή σας και ξέρετε ότι είχα αναφερθεί σε ένα κάπως διαφορετικό πρόβλημα. Μιλούσα για περιοχές όπου καλλιεργούνται γεωργικά προϊόντα, εκτρέφονται ζώα. Είναι ένα πρόβλημα που διαπιστώνεται συχνά από τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, από τους διάφορους συνεταιρισμούς που κάνουν αναλύσεις και βρίσκουν τέτοια προϊόντα όπως τα PCB, τις διοξίνες ε, και μια σειρά άλλων προϊόντων. Ε, λόγω των εκπομπών από τους αποτεφρωτήρες και τις τσιμεντοβιομηχανίες υπάρχουν ε, πολλά προβλήματα όπως είπαμε προηγουμένως σε δύο-τρία διαφορετικά μέρη υπάρχει απόσταση λίγων χιλιόμετρων ανάμεσα σε τέτοιες εγκαταστάσεις, ανάμεσα σε ποτεφρωτήρες ή ε, τις ε, τσιμεντομιομηχανίες και άρα υπάρχει μια, ε, ένας πολλαπλασιασμός των αρνητικών επιπτώσεων και πρόκειται για μονάδες που λειτουργούν εδώ και 60 χρόνια. Ξέρετε, τα ανώτατα όρια δεν είναι απόλυτες τιμές, πρόκειται προς το παρόν για ποσοστά. θα πρέπει να γίνει ανάλυση της ε, λειτουργίας επί σειρά ετών αυτών των ε, μονάδων για να εκτιμηθεί αν, υπάρξει, ε, αν υπάρχει υπέρβαση των οριακών τιμών όπως προτείνονται μέσα στον κανονισμό. Δεν πρόκειται για απαγόρευση της μόλυνσης. Τα κράτη-μέλη απαγορεύουν τη μόλυνση άνω ενός συγκεκριμένου ποσοστού. Λοιπόν, περνάω τώρα στην ερώτησή μου. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν πρόκειται για τυχαία γεγονότα, πρόκειται για ε, περιπτώσεις που παρατηρούνται σε όλη την επικράτεια της ε, χώρας ε, και σας ερωτώ το εξής, δεν κρίνεται ότι θα έπρεπε να διεξάγεται μία ειδική μελέτη για αυτές τις περιοχές όπου υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση αποτεφρωτήρων ε, και μονάδων ε, τσιμεντοβιομηχανίας. Εγώ προέρχομαι από μια περιοχή όπου παράγεται το γνωστό σε όλους μας προσέκο. Καλλιεργούνται τα στέμφυλα για το προσέκο και κατόπιν εξάγεται το προϊόν στην Ευρώπη. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα επώφελες προϊόν ε, προέρχονται από τους λόφους ε, που βρίσκονται κοντά στην Βενετία και από άλλες περιοχές. Τέλος γιατί τα λέω όλα αυτά. Τα κατάλοιπα των ζυζανιοκτώνων. Τα ανώτατα όρια όπως προβλέπονται επιτρέπουν την ε, χρήση κάποιων ζυζανιοκτώνων σε ορισμένα ποσοστά, όμως οι γεωργοί χρησιμοποιούν αυτά τα προϊόντα ε, σε υψηλά ποσοστά ακόμη και αεροσκάφη χρησιμοποιούν για ένα αέριο ψεκασμό για να καλυφθούν όλοι οι αμπελώνες, όλοι οι λόφοι, καταλαβαίνετε, όπου καλλιεργούνται τα στέμφυλα για το προσέκο. Και ανησυχούμε πάρα πολύ στην Ιταλία γιατί τι συμβαίνει. Οι, κάποιοι γεωργοί χρησιμοποιούν αυτά τα παρεστοκτόνα στους αμπελώνες τους Βέβαια οι ίδιοι φορούν στολή, μάσκα κτλ. Και αυτό γίνεται δίπλα ε, σε παιδότοπους, δίπλα σε ευρωφωνηπιακούς σταθμούς, δίπλα σε νηπιαγωγεία. Ε, λοιπόν, στην Ιταλία δεν ε, ε, έχει αναλυφθεί κανένα προληπτικό μέτρο για να προστατευθούν αυτά τα παιδιά. Ξέρω ότι δεν μιλάμε για τρόφιμα και θα μου πείτε ότι είμαι εκτό θέματο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πρόκειται για προϊόντα που θα καταναλωθούν από ανθρώπους, έτσι, γιατί είπαμε τα στέμφυλλα τα χρησιμοποιούμε για το προσέκο που στη συνέχεια πίνουμε. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο ανήσυχοι είμαστε. Ε, σημειώνεται μείωση των αριθμών θανάτου ε, λόγω καρκίνου, ναι μεν, αλλά αυξάνεται ετησίως ο αριθμός αυτών που νοσούν. Λοιπόν, σε όλες τις οικογένειες ε, κάποιος ε, συγγενής ε, πάσχει από καρκίνο. Μήπως θα μπορούσατε να μας δώσετε μία απάντηση για να προστατεύσουμε τους καταναλωτές που... Συγγνώμη, λέει ο κύριο Σλάιτερ, θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο. Αν θυμάμαι καλά τον κανονισμό, ήδη έχουμε απαγορεύσει τώρα τον εναέριο ψεκασμό των παρασιτοκτόνων σε περιοχές που είναι κοντά σε σχολεία και και παιδότοπους. Τέλο πάντων, θα δώσετε εσεί την ερώτηση, αλλά ακού... την απάντηση, αλλά θα ακούσουμε και τι υπόλοιπε ερωτήσει. Ο κύριο ε, Ρώση τώρα. Ευχαριστώ. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η παρουσίαση που μα κάνατε. Όμω ε, έλειπε κάτι σημαντικό. Ποιε είναι οι λύσει. Δεν μιλήσατε για τι λύσει. Μιλήσαμε για την Ασπαρτάμι, για τι 600 μελέτε για... Ε, που αποτελούν πηγή ανησυχία. Ωραία, τι κάνουμε λοιπόν. Περιμένουμε να δημοσιευτούν και άλλε μελέτε. Υπάρχει κάποια θεωρία. Τι περιμένουμε ακριβώ. Έχουμε ένα κανονισμό για την ε, ετικετοθεσία και υιοθετήθηκε αυτός ο κανονισμός και από εμά στην Ολομέλεια. Λοιπόν, καλούνται εκεί τα κράτη-μέλη να επιμείνουν να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα σύμβολα στις ετικέτες που εναποτίθενται στα προϊόντα για τις ε, θερμίδες. Μάλιστα, αυτό το προβλέψαμε. Δηλαδή, εμείς προωθούμε τη δημοσίευση στοιχείων πάνω σε αυτά ε, τα διατροφικά προϊόντα και προαγάγουμε έτσι την ε, χρήση των γλυκαντικών ουσιών ενώ μπορεί να έχουν αυτές οι γλυκαντικές ουσίες όπως η ασπαρτάμι ε, αρνητικές επιπτώσεις. Εγώ το έχω ξαναπεί ενώπιον της Επιτροπής ότι πρόκειται για σκάνδαλο όταν ψηφίζαμε εκείνον τον κανονισμό αλλά δυστυχώς η πλειοψηφία το υπερψήφισε. Επίσης η Coca-Cola Zero λέει ότι αντεδείκνεται για τις εγγύους και για τα ε, παιδιά μέχρι τριών ετών. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια αμφιβολία έτσι, για την ασφάλεια. Λοιπόν, τα κράτη-μέλη θα έπρεπε να χρησιμοποιούν ε, ε, σύμβολα, όχι όμως... Ε, αναδεικνύοντας σε καλύτερα κάποια προϊόντα που ενέχουν γλυκαντικέ ουσίες και να μην αφήνουμε να παρουσιάζονται ω διαιτητικά και υποφελή προϊόντα τώρα. Τα ε, φυτοϊγειονομικά προϊόντα. Κάνουμε τις μελέτες για τα προϊόντα που προέρχονται από τις ε, τρίτες χώρες ε, και όπως είπαν και οι συνάδελφοι υπάρχουν κάποιοι γεωργοί που χρησιμοποιούν κατά κόρον φυτοϊγειονομικά φάρμακα για να αυξήσουμε την παραγωγή της. Μάλιστα, η λύση θα ήταν να μην τα καταναλώνουμε μέσα αυτά τα προϊόντα. Πλην όμως γνωρίζουμε πολύ καλά ότι στην ε, Κίνα χρησιμοποιούνται τοξικά προϊόντα, πολύ πιο επικίνδυνα προϊόντα σε σχέση με την Ευρώπη, πολύ πιο επικίνδυνα και το τονίζω. Μάλιστα, τι κάνει η Ευρώπη από πλευράς ε, ελέγχων. Εγώ ξέρω ότι από μόνη της η Ιταλία για αυτά τα πλαστο... τα παραποιημένα προϊόντα δεν κάνει ιδιαίτερες προσπάθειες για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας και ε, το 40% των παραβάσεων ε, που παρατηρούνται στην Ευρώπη προέρχονται από την Ιταλία γιατί έχουν εντοπιστεί τέτοια προϊόντα στην αγορά μας. Άρα το υπόλοιπο 60% είναι σε άλλες χώρες. Λοιπόν, στο Άμστερνταμ, στο Ρότερνταμ, τι έλεγχοι γίνονται για αυτά τα προϊόντα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι προτίθεται να κάνει για να δώσει μια λύση σε αυτό το πρόβλημα, οι διοξίνες που έχουν εντοπιστεί τώρα. Βεβαίως, βεβαίως οποιαδήποτε και αν είναι η διαδικασία καύσης, εάν δεν προηγηθεί ε, κατάλληλη επεξεργασία του καπνού παράγονται ε, διοξίνες. Οι καυστήρες ε, που λειτουργούν με καυσόξυλα για την παραγωγή ενέργειας δεν δημιουργούν πρόβλημα, κυρίως όταν καίγονται σφαιρίδια, τα «pellets». Ε, εκεί δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με την παραγωγή διοξινών. Αναρωτιέμαι. Φυσικά υπάρχει πρόβλημα. Οπότε, γιατί ε, δεν μας προτείνει κάτι συγκεκριμένο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει να προβλεφθεί απόσυρση αυτής συγκεκριμένη ε, μεθόδου παραγωγής με τα σφαιρίδια. Ε, τώρα, αραβός ή γενετικά τροποποιημένος. Το, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, απεφάνθη. Πρέπει να καταβληθούν αποζημιώσεις στους μελισσοκόμους και στους γεωργούς, μάλιστα. Όμως, θα πρέπει να αποφασίσουμε, να δούμε ε, ποιος έχει δίκιο. Έχει δίκιο το δικαστήριο. Ε, ε, εν τη θα πρέπει να καταβληθούν οι αποζημιώσεις. Καταλαβαίνετε ότι πέρα από την περιγραφή των προβλημάτων θέλω συγκεκριμένε απαντήσει. λέει ο κύριο Λάιτερ, σε σχέση. Όταν σπούδαζα εγώ ε, μηχανικό σε ε, βιομηχανίε, είδαμε ότι η καύση σχετίζεται με την μέθοδο παραγωγής, με τη μέθοδο καθαρισμού κτλ. Και σε ολόκληρη τη Σουηδία, να σας πω ότι η χειρότερη μόλυνση είναι σε, μία, σε ένα μικρό χωριό, σε μία κομμόπολη που χρησιμοποιούν όλοι καυσόξυλα. Καταλαβαίνετε ότι η ρήπανση μπορεί να προέλθει από μικρής κλίμακας ή μεγάλης κλίμακας ε, μονάδες. Καλ Χάινσε, θέλεις το λόγο. Όχι. Ακούμε την απάντησή σα Λέβα. Μάλιστα, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Να ξεκινήσω με αυτά που αναφέρατε για την ενδεχόμενη μόλυνση κατά το παρελθόν κοντά σε βιομηχανικά εργοστάσια. Διοξίνες ή ενδεχομένως και άλλα χημικά, συστατικά και άλλες χημικές ουσίες. Πρώτο σχόλιο, θα ήθελα να σας πω ότι για τους μολυντές που έχουν ρυθμιστεί από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, είναι σαφές ότι υπάρχουν ανώτατα επίπεδα. Αν δεν γίνονται σεβαστά το προϊόν, πολύ απλά δεν διατίθεται στην αγορά. Αυτό ως πρώτο σχόλιο. Ύστερα, μια άλλη πτυχή που τίθεται είναι είναι ότι μπορεί να υπάρχουν περιοχές κοντά σε παλαιά εργοστάσια και ενδεχομένως στο παρελθόν δεν ήταν τόσο καλή η προστασία όπως αυτή που έχουμε σήμερα, γιατί για παράδειγμα έχουν εισαχθεί φίλτρα υποχρεωτικά για να αποφευχθεί η μόλυνση στις περιοχές της γειτονικέ του εργοστασίου. Άρα, στο παρελθόν μπορεί να υπήρχαν τέτοιες εκπομπές οι οποίες να είχαν προκαλέσει υψηλή μόλυνση. Και μπορεί να υπάρχουν και αγροτικές εκμεταλλεύσεις κοντά στις περιοχές αυτές. Αλλά θεωρώ ότι το πρόβλημα αυτό δεν εντάσσεται στο πεδίο της εντολής μας. Ε, αυτό εναπόκειται στους υπεύθυνους στο εθνικό και τοπικό επίπεδο. Αυτοί θα πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτή τη δύσκολη κατάσταση σε ό,τι αφορά τον περίγυρο ε, των παλαιών εργοστασίων, όπου υπάρχει ενδεχομένως ε, μολυσμένο έδαφος, ε, όπου υπάρχουν γεωργικές εκμεταλλεύσεις, εκτροφές και ενδεχομένως να υπάρχουν προβλήματα από το υψηλό επίπεδο μόλυνσης, το οποίο ενδεχομένως να οδηγήσει σε υψηλή παρουσία μολυντών. Αυτό όμως δεν αποτελεί ένα αντικείμενο στο το οποίο εντάσσεται στο πεδίο αρμοδιότητας της ΕΦΣΑ. Αλλά για τις διοξίνες έχουν τεθεί άνω τα επίπεδα ε, στην νομοθεσία, τα οποία πρέπει να γίνονται σεβαστά για τα ζυζανιοκτώνα, τα παραστακτόνο αν κατάλαβα σωστά την ερώτηση, αναφερθήκατε σε συγκεκριμένες πρακτικές σε μια περιοχή όπου καλλιεργούνται αμπελώνες για το προσέκο, αλλά φαντάζομαι ότι συμβαίνει και αλλού αυτό. Αναφερθήκατε στο γεγονός ότι τα παραστοκτόνα ενδεχομένως να ψεκάζονται με τέτοιο τρόπο που να έχουν ενδεχομένως αντίκτυπο στους κατοίκους της περιοχής ή και στους εργαζόμενους. Εμείς ε, αξιολογούμε κατά την αξιολόγηση κινδύνου όχι μόνο τον αντίκτυπο στην υγεία του καταναλωτή αλλά και τον αντίκτυπο στην υγεία του αγρότη, του εργαζόμενου αλλά και στην υγεία των κατοίκων, των περιοίκων. και άρα αυτό αποτελεί σημαντικό τμήμα της δουλειάς μας. Και αυτή η δουλειά καταλήγει σε κάποια μέτρα διαχείρισης κινδύνου. Άρα, όταν κάποια παρασυντοκτόνα διατίθενται στην αγορά, υπάρχουν συστάσεις. Οι βέλτιστες, αν θέλετε, αγροτικές πρακτικές, οι οποίες διασφαλίζουν ότι ο τρόπος χρήσης των παρασυντοκτόνων δεν θα επηρεάσει αρνητικά όσους ζουν κοντά στην περιοχή αυτή. Είτε πρόκειται για σχολεία, είτε πρόκειται για κόσμο που ζει απλά στην περιοχή. Δεν είμαι σίγουρη αν κατάλαβα σωστά την ερώτηση. Για την Ασπαρτάμι. να πω ότι λυπάμαι αν δεν ήμουν αρκετά σαφής. Έχουμε λάβει 600 έρευνες, μελέτες και θα προβούμε σε μια αξιολόγηση κινδύνου. Το έργο αυτό είναι σημαντικό. Σας είπα ότι πρόκειται να πάρει χρόνο, γιατί πρόκειται για με πλήρη εκτίμηση, αξιολόγηση κινδύνου και επίσης θέλουμε να συμπράξει και η επιστημονική κοινότητα εντός και εκτός Ευρώπης, γιατί ξέρουμε ότι το θέμα είναι αμφιλεγόμενο. Δεν θα έλεγα ότι το θέμα αυτό είναι καταπήγον. Αναφέρθηκα προηγουμένως στην παρουσίασή μου σε πολλά θέματα τα οποία είναι καταπήγοντα και που θα πρέπει να θα αντιμετωπίσουμε άμεσα, για παράδειγμα, χημική μόλυνση τροφίμων κτλ. Εδώ δεν υπάρχει καταπήγον χαρακτήρα. Είναι σημαντικό να γίνει σωστή δουλειά. Και γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι αξίζουν οι επιστήμονές μας κάποιους μήνε προκειμένου να εργαστούν σωστά. Εισάγουμε πολλά φυτά από άλλες ε, χώρες ε, και αυτό που αποτελεί η πρόθεσή μας είναι να εισάγουμε το φυτό και όχι την νόσο, όχι τη μόλυνση. Ζητήθηκε από, ε, από την έψα να κάνει μία έρευνα σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση κινδύνου για τέτοιους ε, παράγοντες μόλυνσης, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι δεν πρόκειται να εισάγουμε φυτά τα οποία θα προκαλέσουν προβλήματα. Φυσικά υπάρχει και ένα σημαντικό ρόλο ε, και από πλευρά Επιτροπή και από πλευρά κρατών μελών που θα πρέπει να διαδραματίσουν για να διασφαλίσουν ότι η νομοθεσία σε ό,τι αφορά τα φυτά τα οποία εισάγονται στην επικράτεια της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν επιβλαβείς οργανισμούς που μπορούν να βλάψουν την γεωργία μας. Αλλά αυτό είναι δουλειά των κρατών μελών και της Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος και προφανώς πρόβλεψα το μέλλον γιατί τώρα ζητάει το λόγο Καν Χάιντς Φλόρενς. Ναι, πάντα είμαι σχετικά αργός, Πρόεδρε μια διαφορετική ερώτηση και δεν ξέρω αν έχετε θίξει το θέμα αυτό γιατί είχα Επιτροπή Συνδιαλλαγής προηγουμένως. Ακούω συχνά ότι στις επιτροπές σας, την ΕΦΣΑ, στις επιστημονικές επιτροπές, υπάρχουν φήμες ότι υπάρχουν πολλοί εμπειρογνώμονε οι οποίοι προασπίζουν συγκεκριμένα συμφέροντα. Είχα κάνει και μια συγκεκριμένη εκστρατεία. Το πρόβλημα αυτό επιλύθηκε ή βρίσκεστε σε μια φάση αντιμετώπισης του προβλήματος. Νομίζω ότι το θέμα αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και αν θα μπορούσατε παρακαλώ να μου απαντήσετε εν συντομία. Ο Πρόεδρος, ναι, το αναφέραμε αυτό το θέμα της σύγκρουσης συμφέροντων. Ίσως όμως, αν θέλετε, να αναφερθώ στο θέμα των παρασυντοκτώνων. Οι εργαζόμενοι προστατεύονται. Μπορεί να υπάρξει περαιτέρω περιορισμός της χρήσης ε, λόγω λανθασμένης διαχείρισης, ε, λόγω λανθασμένης χρήσης που δεν προστατεύει την, ε, τους περίοικους. Έχετε αρμοδιότητα να περιορίσετε τη χρήση των ε, παρασιτεκτόνων επειδή δεν χρησιμοποιούνται σωστά, ακόμα και αν δεν έχουν επίδραση στα τρόφιμα. Σας ευχαριστώ. Κοιτάξτε, του χρόνου, αν δεν κάνω λάθος, θα μπορέσουμε να δημοσιεύσουμε μία μεθοδολογία η οποία θα βελτιώσει την αξιολόγηση κινδύνου σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπο των παραστακτώνων στους εργαζόμενους, στους περίοικους. Άρα, βρισκόμαστε σε φάση αξιολόγησης του θέματος αυτού και καταρτίζουμε πολλά σχετικά έγγραφα και του χρόνου θα δημοσιεύσουμε σχετική μελέτη για να ληφθεί υπόψη καλύτερα ο αντίκτυπος. Και θα ήθελα επίσης να αναφέρω, επειδή ξέρω ότι αυτό σας ενδιαφέρει εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ότι ενδιαφέρει και πολλούς Ευρωπαίους πολίτες, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας ζήτησε να βελτιώσουμε την μελέτη αντικτύπου, την αξιολόγηση κινδύνου σε ό,τι αφορά την χρήση παραστοκτώνων για τις μέλισσες. Του χρόνου λοιπόν θα δημοσιευτούν τα έγγραφα αυτά. Πολύ σημαντική δουλειά και αυτή σε ό,τι αφορά την δήλωση συμφερόντων για να διαβεβαιώσω τον κύριο Φλόρεντς ότι όντως ε, αντιμετωπίζουμε το θέμα αυτό. Οποτεδήποτε διατυπώνεται κριτική, ανησυχία σε ό,τι αφορά ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων για τους εμπειρογνώμονές μας, ε, απαντούμε. Δεν λέω ότι πείθουμε πάντα, αλλά τουλάχιστον δίνουμε μία απάντηση. Και λαμβάνουμε υπόψη και τον τρόπο που γίνεται αντιληπτό το έργο μας σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των κανόνων αυτών. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Είμαι βέβαιος ότι θα το συζητήσουμε και του χρόνου το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ που ήρθατε λοιπόν εδώ στην Επιτροπή μας και σας εύχομαι καλή τύχη, καλή συνέχεια και έτσι ολοκληρώνουμε το σημείο αυτό στην ημερήσια διάταξη. Όπως σας είπα και προηγουμένως, ε, το επόμενο θέμα θα ξεκινήσει στις 5 γιατί τότε θα καταφτάσουν οι αρμόδιοι συνάδελφοι. Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα λοιπόν και ξαναξεκινάμε στις 5.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 Uh, let's subject and Συνεχίζουμε. Έχουμε τον εισηγητή μας, τον κύριο Γιώκενσον, που θα συζητήσουμε μαζί του εξαγωγές και εξαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων. Τα χημικά είναι το αγαπημένο μου θέμα, ε, οπότε σας ακούμε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω παρουσιάζοντάς σας ε, κάπως το θέμα. Πρόκειται για την σύμβαση του Ρότερνταμ που προβλέπει ανταλλαγές πληροφοριών όσον αφορά εισαγωγές και εξαγωγές επικίνδυνες χημικών προϊόντων. Όταν εξάγονται ε, τέτοια προϊόντα από ένα μέλος της σύμβασης σε ένα άλλο μέλος της σύμβασης. Πρόκειται για ένα μηχανισμό ο οποίος διασφαλίζει ότι οι χώρες που εξάγουν ε, τέτοια προϊόντα παίρνουν ρητά την συμφωνία από τη χώρα στην οποία θα εξαχθεί το προϊόν ότι όντως συμφωνούν να εισάγουν το προϊόν αυτό. Υπάρχουν τάρτρα τα οποία προβλέπουν τα ζυζανοκτόνια και τα χημικά. Ορισμένα από αυτά απαγορεύονται ρητά, για λόγους είτε περιβάλλοντος ή για άλλους. Τώρα, Αν δούμε τη συγκεκριμένη πρόταση που έχουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτα απ' όλα επιτρέψτε μου να σας πω δύο λόγια για τα κάπως πιο τεχνικά ζητήματα και μετά θα περάσουμε στα πιο πολιτικά. Όπου εκεί διαφωνώ εν μέρη με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έρχομαι λοιπόν πρώτα στα τεχνικά όπως είπαμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να διευκρινίσει κάποιους ε, κανονισμούς προκειμένου να τους ευθυγραμμίσει με άλλη νομοθεσία που έχει υιοθετηθεί από τότε που τέθηκε σε εφαρμογή ο... Ε, η σύμβαση αυτή. Εδώ συμφωνώ, αλλά προτείνει επίσης κάτι για την εφαρμογή του κανονισμού. Εδώ χρειαζόμαστε υψηλού επίπεδου εμπεριματοσύνη και δεν πιστεύω ότι πρέπει να βιαστούμε. Έρχομαι όμως στα κάπως πιο πολιτικά ζητήματα. Το πιο προβληματικό θέμα της πρότασης της Επιτροπής είναι ότι η Επιτροπή αποδυναμώνει τον ε, κανονισμό όσον αφορά την ε, σύμφωνη γνώμη. Λέει δηλαδή ότι οι εξαγωγείς που δεν έχουν πάρει μέσα σε 60 μέρες απάντηση από το κράτος μέλος το οποίο θα εξάγουν το προϊόν τους, τότε να μπορούν να κάνουν την εξαγωγή αυτή. Με την πρόταση της Επιτροπής θα προσθεθεί ένα άρθρο 14 το οποίο θα επιτρέπει, όπως σας είπα, εφόσον έχει χρησιμοποιηθεί ε, προηγουμένως το προϊόν αυτό, εφόσον έχει εγκριθεί τα τελευταία πέντε χρόνια και δεν υπάρχει τίποτα που να αντιβαίνει στην ε, εισαγωγή αυτή, να μπορούν να κάνουν την ε, εξαγωγή τους στην χώρα που θέλουν να εξάγουν. Αν δεν έχουν πάρει απάντηση, εντό 60 ημερών μπορούν να εξαγάγουν το χημικό προϊόν, εφόσον υπάρχει απόδειξη ότι το χημικό προϊόν έχει αποτελέσει αντικείμενο έγκριση, χορήγηση άδεια ή καταχώρηση στη χώρα εξαγωγή. Υπάρχει το παράρτημα 1, τα σημεία 2 και 3, που λένε μέχρι τώρα ότι δεν μπορεί να γίνει η εξαγωγή αυτή επειδή δεν υπάρχει απάντηση από την χώρα εισαγωγής. Στην έκθεσή μου φαίνεται, τι είναι αυτό που πιστεύω εγώ, ότι δεν είναι καλή ιδέα να αλλάξουν αυτά, γιατί για ποια χημικά πρόκειται εδώ. Αναφέρονται στο παράρτημα 1, σημεία 2 και 3. Είναι χημικά τα οποία είτε είναι απαγορευμένα είτε χρησιμοποιούνται πάρα πολύ λίγο. Πολύ περιορισμένη χρήση λοιπόν ή απαγόρευση. Οπότε δεν βλέπω γιατί για εμπορικού λόγους να επιτρέψουμε παρέκκληση για τέτοιου είδους χημικά. Αν μια χώρα σε 60 μέρες δεν έχει απαντήσει, μπορεί αυτό να συμβαίνει για διάφορους λόγους. Σύμφωνα με την Επιτροπή δεν απαντάει επειδή θεωρούν ότι δεν χρειάζεται. Μπορεί όμως να σημαίνει και κάτι άλλο. Μπορεί να υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Επειδή δεν έχουν τους πόρους, τους δικητικούς να ασχοληθούν με την απάντηση αυτή. Δεν σημαίνει ότι το επιτρέπουν κιόλα. Αν μάλιστα δούμε τα επίσημα στοιχεία που έχουμε από τα Ηνωμένα Έθνη, εκτιμούν ότι κάθε χρόνο 47 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους από τέτοια χημικά. 47.000 άνθρωποι, σχεδόν 5.000. Εννοείται και πολύ περισσότεροι έρχονται να με ασθένειε ή αναπτύσσουν κάποια σύνδρομα ή αρρωσταίνουν εξαιτία της ε, χρήσης τέτοιων χημικών. Οπότε πρέπει να προστατεύουμε όσο μπορούμε περισσότερο τους ανθρώπους και όχι για εμπορικούς λόγους να επιτρέπουμε τις εξαγωγές αυτές. Έπειτα, η ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον είναι ε, τα στοιχεία, οι όροι που περιλαμβάνει η σύμβαση του Ρότερνταμ. Ότι αυτά θέλουμε να προστατεύσουμε. Και εγώ δεν βλέπω να προστατεύονται αυτά με παρετέρω παρεκκλήσεις. Συνεπώ, πιστεύω ότι πρέπει να πάμε προς την αντίθετη κατεύθυνση. Πιστεύω ότι πρέπει να ενισχύσουμε τον κανονισμό ακόμα περισσότερο, ώστε να είναι ακόμα πιο δύσκολο να υπάρξει παρέκκληση όταν μιλάμε για ιδιαίτερα επικίνδυνες χημικές ουσίες. Αναγνωρίζω ότι μπορεί να υπάρχουν πραγματικά εξαιρέσεις και να μπορέσουμε ενδεχομένω να δεχτούμε κάποια παρέκκληση, αλλά γενικά όχι, να μην υπάρχουν τέτοιες παρεκκλήσεις. Δεύτερον, που είναι επίσης πολιτικό θέμα, είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει πως μόνο η Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση στη Σύμβαση. Όμως, εάν ο κανονισμός βασιζόταν καθαρά σε εμπορικέ βάσει θα είχε νόημα, γιατί πραγματικά μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί ε, προ τα έξω για εμπορικά θέματα να εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμω βασίζεται και σε εμπορική ε, νομική βάση, αλλά και σε περιβαλλοντική νομική βάση. Και θυμόσαστε που είχαμε στο δικαστήριο το 2006. Έπειτα πρόκειται για επιμερισμένη ευθύνη κρατών μελών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε και τα κρατη και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν την ευθύνη και άρα πρέπει να εκπροσωπούνται στη σύμβαση. Δεν συμφωνώ δηλαδή να είναι μόνο η Επιτροπή. Τέλος, το πιο σημαντικό είναι το κατά πόσο πρέπει να επιτρέψουμε ή όχι στους εξαγωγείς εφόσον δεν έχουν πάρει απάντηση μέσα σε κάποιο χρονικό διάστημα να συνεχίσουν με την εξαγωγή τους αν μπορούν να αποδείξουν ότι τα χημικά αυτά έχουν εξαχθεί κατά το παρελθόν ε, στην ε, χώρα εισαγωγή. Εγώ δεν συμφωνώ. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να επιτρέπεται κάτι τέτοιο. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνει ακόμα πιο αυστηρός ο κανονισμός για να υπάρχουν όλο και λιγότερε δυνατότητε να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. εσύ εδώ πέρα εκπροσωπείς ε, την συγκέντρια Μακίνησε. Ευχαριστώ. Δυστυχώ δεν μπορεί να παρευρεθεί η κυρία Μακίνη και γι' αυτό με παρακάλεσε να παρουσιάσω τι ε, απόψει τη και τι απόψει τη ομάδα μα για την πρόταση αυτή. Σε μεγάλο βαθμό συμφωνούμε με τον Νταν Γιούργενσεν και με την ανάλυση που έκανε, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά με τα τμήματα εκείνα τα οποία παρουσίασε για την συμμετοχή των κρατών μελών η νομική βάση είναι σαφής. Και θεωρούμε ότι και τα κράτη-μέλη πέρα από την Επιτροπή θα πρέπει να συμμετέχουν στην άλλη διαδικασία γιατί όπως αναφέρθηκε πρόκειται για θέμα κοινή αρμοδιότητας και σε ό,τι αφορά τη μεταφορά αρμοδιοτήτων ε, από τα κοινά αρνητικά κέντρα στα πλαίσια της ε, ε, ΕΚΑ είναι σημαντική και σε ό,τι αφορά τη διαδικασία επιτροπολογίας, αυτά που αναφέρει ο εισηγητής, μας βρίσκουν σύμφωνους. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον συνάδελφο Γιώργενσεν να διευκρινίσει λίγο πιο καλά τους λόγους τους, για του οποίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβη στη διατύπωση των εξαιρέσεων αυτών σε ό,τι αφορά την πρώτερη συγκατάθεση και σε ό,τι αφορά την μη τήρηση του χρονικού πλαισίου. Μήπως ανοίγουμε μία ε, πόρτα μέσω της οποίας μπορούν να εξαχθούν ε, επικίνδυνες χημικές ουσίες χωρίς τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Νομίζω όμως ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπή έχει κάποια ουσία και θα πρέπει να διεξάγουμε κάποια συζήτηση για το πώς μπορούμε να περιορίσουμε για να σε ό,τι αφορά μάλλον την δυνατότητα να μην ανοίξουν παραθυράκια, δεν συμφωνούμε απόλυτα. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια αν ε, δεν έχουν γίνει ε, εγκαίρως οι αιτήσει για έγκριση. Θα θέλαμε επίσης να προτείνουμε ιδιαίτερο σε ό,τι αφορά τα διπλά πρότυπα αν μια χημική ουσία επιτρέπεται στην κοινότητα και μπορεί να τύχει επεξεργασία. θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι γίνεται σε άλλες χώρες. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να έχουμε ανταγωνιστικό μείον έκτημα. Θα πρέπει να ισχύουν οι ίδιοι όροι για όλους. Νομίζω ότι υπάρχουν οικονομικοί λόγοι για τον περιορισμό τέτοιων απαγορεύσεων, γιατί ιδάλλως ποια θα είναι η συνέπεια τα χημικές αυτές ουσίες θα προέρχονται από άλλες τρίτες χώρες και θα βρεθεί σε μενεκτική θέση η βιομηχανία μας. Άρα νομίζω ότι θα πρέπει να αναφερθούμε στο θέμα των τρίτων χωρών και στις χημικές ουσίες, να μην δεν έχει νόημα να απαιτούμε πιο αυστηρέ προδιαγραφέ από τρίτε χώρε από ό,τι στο εσωτερικό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, Όπω σα είπα, η πρόταση του Νταν Γιώργενσεν για την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρήζει περαιτέρω συζήτηση για τον περιορισμό των ε, δυνατοτήτων παράβλεψη των κανονισμών, αλλά χωρί ολική απαγόρευση. Σα ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρο και επόμενη σκιώδη, η Όλγα Κρέμερ. Ο Όλγα Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι συμφωνώ με αυτά που είπαν οι συνάδελφοι. Δεν έχω να προσθέσω κάτι ιδιαίτερο. Νομίζω ότι σε Γενικέ γραμμέ θα πρέπει να ακολουθήσουμε τι προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά διευκρινήσει που χρειάζονται και για τη συμπερίληψη του, της ΕΚΑ και τι προσαρμογέ σε ό,τι αφορά τη συνθήκη της Λισαβόνας. Να μην επαναλαμβάνω όμω αυτά που ακούσαμε. Να σα προειδοποιήσω μόνο να μην δοθεί υπερβολικά πολιτικός χαρακτήρας στο, ε, στο θέμα αυτό. Ασχολήθηκα πολύ με το θέμα αυτό το Σαββατοκυριακό. Η δυνατότητα παρέκκλησης από αυτά που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι τόσο στενές που δεν θεωρώ απαραίτητα ότι θα πρέπει να, το, να δώσουμε συνέχεια. Μας ανέφερε τη σχετική μελέτη ο Νταν για τα 47.000 άτομα που χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο επειδή έρχονται σε επαφή με διάφορες χημικές ουσίες. Νομίζω ότι η σχετική μελέτη του ΟΙΕ είναι πολύ πιο γενική. Έχει άλλη βάση και θα μπορούσαμε να θέσουμε και το αντίθετο ερώτημα. Πόσα άτομα πεθαίνουν από υποστηρισμό γιατί περιορίζεται η πρόσβαση στα φυτικά μέσα. Νομίζω λοιπόν ότι είναι περιττό να μπλέξουμε αυτό το θέμα στην συνηθισμένη συζήτηση για τις χημικές ουσίες. Νομίζω, το είπε και ο κύριος ε, Ζέιμπερ, ότι θα πρέπει να λογιστούμε και τις συνέπειες. Ε, μιλάμε ε, για την πρακτική εφαρμογή των εμπορικών μηχανισμών. Αν κλείσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτές τις διόδους ε, Πολύ απλά θα λαμβάνουμε τα χημικά αυτά από άλλους παραγωγούς οι οποίοι δεν θα τηρούν τις προδιαγραφές αυτές. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει πολύ προσεκτικά να σκεφτούμε κατά πόσον μπορούμε να εισαγάγουμε τους ίδιους όρους όπως και για τα μέτρα προστασίας των ε, φυτών για τα διπλά πρότυπα. Νομίζω ότι ε, όλα αυτά περιπλέκουν περαιτέρω τη συζήτηση. Να πω λοιπόν ότι επί της ουσίας ε, μας ε, βρίσκει σύμφωνος η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νομίζω ότι προσαρμόζει την νομοθεσία αυτή στην πραγματικότητα. Thank you. And Σας ευχαριστώ. Να Ρόσμπαχ, αντικαθιστά την Τζούδιθ Κάρλιν, παρακαλώ. Ναι, Όντως, μου ζήτησε τουλάχιστον διαβάσω τη δήλωσή της, τη θέση της. Θέλει να ευχαριστήσει τον εισηγητή για την έκθεση, να υποστηρίξει τις τροπολογίες του, όπου επαναφέρει διατύπωση από τον αρχικό κανονισμό του 2008 για το άρθρο 5. Συμμερίζεται δηλαδή την άποψή του ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να διαθέτουν τη διακριτική του ευχαίρεια κατά την εφαρμογή τη σύμβαση ε, του Ρότερνταμ. Εμφανιστεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τι εισηγήσει τη και εν γέννη υποστηρίζει το νέο σχέδιο του κανονισμού σίγμα 1 ε, με τους ορισμούς, ε, τους ε, κανόνες βάσει του κανονισμού CLP για να αυξηθεί η συμμετοχή της ΕΤΑ και θέλει να στηρίξει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με τη διαδικασία ΠΙΚ ε, για τις ε, χώρες που εισάγουν ε, βάσει του άρθρου 3.7 Διευκρινίζει βεβαίω ότι χρειάζεται περαιτέρω αναθεώρηση τη διατύπωση. Όμω με την ιδιότητα του συνομοθέτη, το Κοινοβούλιο δεν θα πρέπει να παραβιάσει τις αρχές της συμβάσης του Ρότερνταμ και ούτε και να εισαγάγει με τις διατάξεις περί τη γραφειοκρατία. Είναι λοιπόν σχετικά ικανοποιημένη όπως βλέπετε. Ευχαριστώ, λέει ο κύριο Σλέτερ. Τώρα με την ιδιότητα του Σκιώδους από πλευράς Πρασίνων θα πάρω και εγώ το λόγο. Ευχαριστούμε και εμείς τον εισηγητή για την πρότασή του. Είναι πολύ καλή. Θα θέλαμε επίσης οι προτάσεις σας να ενισχύσουν τον κανονισμό και όχι να δημιουργήσουν ε, περαιτέρω εξαιρέσεις. Δεν μας ικανοποιεί η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με αυτή τη λογική ότι εφόσον έχει τεθεί σε εμπορία νωρίτερα μπορεί να συνεχίσει η εμπορία λόγω και μόνο αυτού. Διότι όταν ένα εξαγωγέας ε, πει ότι αφού οι ανταγωνιστέ μου το πουλάνε, γιατί να μην συνεχίσω κι εγώ εσάι να πουλάω αυτό το προϊόν. Όχι, δεν μπορεί αυτό να συνιστά ικανοποιητικό κριτήριο. Ο πρωταρχικός στόχος ε, του κανονισμού είναι αυτό το prior informed consent που λέμε. Ε, δηλαδή, συγκατάθεση συνέχιση μάλλον μετά από ενημέρωση. Δηλαδή θα πρέπει κάποιο να έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί πρώτα για τη χημική ουσία και να αποφασίσει μετά. Και τι σημαίνει consent, ε, ε, συγκατάθεση. Όχι υποθέτουμε ότι όλα Λαβέν Σίος επειδή κυκλοφορούσε ένα προϊόν. Και νομίζω ότι η πρόταση του Ντάν ακολουθεί αυτή τη λογική που μόλις εξέθεσα και άρα μας ικανοποιεί. Ξέρετε, δεν πρέπει να κάνουμε στου άλλου αυτά που δεν θέλουν να μα κάνουν. Ε, είναι σημαντικό. Και αν απαγορεύσουμε κάτι και στη συνέχεια προβλέψουμε εξαιρέσει για τη διευκόλυνση του εμπορίου, νομίζω ότι το παρακάνουμε. Θα έπρεπε να εμείνουμε σε αυτή τη λογική τη συνέχιση μετά από ενημέρωση στο μέτρο του δυνατού και να ελεγχιστοποιήσουμε τον αριθμό των εξαιρέσεων. Αυτή είναι η άποψή μου ε, ως σκιώδης εισηγητή. Δεν έχει ζητήσει κανένας άλλος το λόγο. Ο Μπιόν Χάνσον είναι εδώ. Α, η... Άστιτ Σόμακερ από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Αντικαθιστώ ε, τον συνάδελφο. Ε, σας ευχαριστώ που εργαστήκατε ταχύτατα σε αυτό το φάκελο. Σας ευχαριστούμε που υποστηρίξατε το σχέδιο των νέων προτάσεων σε μεγάλο βαθμό που καταθέσαμε. Θα ήθελα να αρχίσω με αυτή την ελή αναφιλεγόμενη παράγραφο, δηλαδή η τροποποίηση της ε, διαδικασίας PIC. Λοιπόν, από τη δική μας οπτική γωνία είναι σημαντικό να πούμε ότι ο κανονισμός ε, ΠΙΚ ε, ήδη υπερβαίνει σε πολλά σημεία τη σύμβαση του Ρότερνταμ, κυρίως για τη διαδικασία συνέχισης μετά από ενημέρωση που εφαρμόζεται σε 106 χημικές ουσίες αυτή τη στιγμή, σε αντίθεση με τις 46 που καλύπτει η σύμβαση του Ρότερνταμ. Επίσης θα ήθελα να διευκρινίσω ότι με αυτό το νέο σχέδιο πρότασης ε, δεν είχαμε ουδόλως την πρόθεση να διαταράξουμε την ισορροπία που ευρέθη το 2008 ανάμεσα στα συμφέροντα ε, των ευρωπαϊκών παραγωγών χημικών ουσιών και εξαγωγείων αυτών ε, και την προστασία του περιβάλλοντος από την άλλη πλευρά, δηλαδή την προστασία από τη χημική ρήπανση. Τρία χρόνια έχουν περάσει από τη θέση σε ισχύ. Κανονικά δεν θα είχαμε επανέλθει τόσο σύντομα για να αναθεωρήσουμε το νομοθέτημα, όμως λόγω των αλλαγών στη δίκη Λισαβόνας, ε, λόγω της ε, προσαρμογής για τη διαδικασία ταξινόμησης και τικετοθεσίας, να είμαστε θα πρέπει να επανεξετάσουμε το άρθρο 14 και να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτή η ισορροπία του 2008 λειτουργεί αισίως. Επίσης, σε 30% των περιστώσεων διαπιστώσαμε και παρά τις προσπάθειες που έκανε είτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είτε η διοριστήσα εθνική αρχή, δεν λαμβάνουμε απάντηση από την χώρα που εισάγει τα προϊόντα. Περιμένουμε μήνες και χρόνια ορισμένες φορές ε, για την απάντηση. Προσπαθούμε να διερευνήσουμε τους λόγου και συμφωνούμε με τον κύριο Γιώργενσεν ότι ενίοτε είναι έλλειψη δυνατότητας ε, ε, για να απαντήσουν όμως χρησιμοποιούμε και το δίκτυο της σύμβασης του Ρότερντον, το διεθνές δίκτυο, για να διερευνήσουμε την υπόθεση. Γιατί λοιπόν δεν λαμβάνουμε τις απαντήσεις ε, και ανακαλύψαμε ότι ε, στις πλήστες περιπτώσεις η διοριστή σε Εθνική Αρχή δεν κατανοεί καν γιατί πρέπει να απαντήσει, γιατί πρέπει να δώσει πληροφορίες για τις χημικές ουσίες εφόσον δεν καλύπτεται από τη σύμβαση για την οποία τόσο αγωνίστηκαν κτλ. Οπότε δεν είναι προστασία στις αναπτυσσόμενες χώρες ε, το θέμα είναι Ευρωπαίος εξαγωγίας ε, που έχει τον ανταγωνισμό από τις τρίτες χώρες για την εξαγωγή της ίδιας ε, χημικής ουσίας προς την ίδια αναπτυσσόμενη χώρα. Έτσι σκέφτεται και υπό το φως αυτών των εμπειριών και παρότι επιθυμούμε να διατηρηθεί η ισορροπία, κρίναμε ότι ήταν σκόπιμο να εισαγάγουμε μια περιορισμένη περαιτέρω δυνατότητα και το τονίζω ότι θα γίνει αυτό σε προσωρινή βάση για τις περιπτώσεις ε, όπου Υπάρχει τεκμηρίωση από επίσημες πηγές που καταδεικνύει ότι έχει εισαχθεί το χημικό προϊόν και έχει χρησιμοποιηθεί τα τελευταία πέντε χρόνια. Δεν έχει γίνει καμία προσφυγή, δεν έχει δοθεί απάντηση για δύο μήνε κτλ. κτλ. Όλο το άρθρο δηλαδή. Και οι εξαγωγεί ε, τότε θα μπορούσαν ε, για μια μεταβατική 12 μήνη περίοδο και αναμένοντα την αίτηση να προβούν στη θέση εμπορία του προϊόντος. Ε, αναμένουμε βεβαίω ε, περαιτέρω διευκρινήσει από τρίτε χώρε που αναλαμβάνουν τέτοια μέτρα. Συνοψίζοντα, ε, είναι μια περιορισμένη απόκληση που τελεί υπό όρου. δεν αναταράσουμε, διαταράσουμε μάλλον σε τίποτα την ισορροπία του 2008. Και εφόσον έχω το λόγο, θα ήθελα εντάχει να σχολιάσω και άλλε δύο τροπολογίε. Υπάρχει παρανόηση κατά τη γνώμη σε σχέση με την εξωτερική εκπροσώπηση. Προτείνουμε την διαγραφή της παραγράφου 1 του άρθρου 5 για τον απλό λόγο ότι το θέμα της εξωτερικής εκπροσώπησης ε, τώρα ρυθμίζεται στην ε, συνθήκη λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και δεν χρειάζεται περαιτέρω διατύπωση υπερισχύει η συνθήκη και φυσικά τα κράτη-μέλη σε τομείς αρμοδιότητός τους εκπροσωπούν αυτούς η πρότασή μα σημαίνει αποφυγή ιονή συγκρούσεων ανάμεσα στο δευτερογενές δίκαιο και τις συνθήκες. Ε, τέλος, ε, ένα λίαν τεχνικό θέμα που δεν σχολίασε καθόλου ο κύριος Γιώργενσεν, εγώ παρόλα αυτά θα ήθελα να αναφερθώ. Ε, μας ανησυχεί η τροπολογία υπαριθμών 4. Ο εισηγητής... Ε, ε, θα αποδυναμώσει την προστασία των ε, αναπτυσσόμενων ε, χωρών. Ποιο είναι το πρόβλημα με την τροπολογία. Οι χώρες που εισάγουν θα έχουν μία κοινοποίηση για όλες τις εξαγωγές, ε, για, όλα, για όλες τις σύνθετες ουσίες που εμπεριέχουν αυτή την χημική ε, ουσία. Ε, δηλαδή δεν θα ενημερωθούν για διάφορες παρτίδες που ενέχουν αυτή την χημική ουσία με διαφορετική όμως εμπορική ονομασία. Ε, και αυτό ε, αναιρεί τα όσα είπαμε για το μητρό και τις εμπορικές ονομασίες ε, των χημικών ουσιών. Λοιπόν, ευχαριστώ τον εισηγητή, ευχαριστώ και όλου του συναδέλφου για τα σχόλιά του και είμαστε στη διάθεσή σα. Ευχαριστούμε κύριο Σουμάχηλο, κύριο Σλάιτερ. Τώρα ο κύριο Τσίμερ, ο θα πάρει πάλι το λόγο. Ένα λεπτό, να κάνω μια ερώτηση θα ήθελα στην Επιτροπή πριν δώσω τις απαντήσεις προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για την τροπολογία 4 μπορούμε να το συζητήσουμε και διεξοδικότερα. μάλλον δίκαιο έχετε και θα χρειαστεί να ανασυντάξω την τροπολογία. Όμως, ε, σχετικά με την διαδικασία συνέχισης μετά από ενημέρωση, ε, μάλλον έχετε δίκιο όταν λέτε ότι κάποιες χώρες δεν απαντούν διότι δεν μπορούν. Ε, όμως, ταυτόχρονα λέτε ότι αν εμείς δεχτούμε την πρότασή σας ε, θα περιέλθουμε στην εξή κατάσταση. Η Ένωση θα αρχίσει να εξάγει χημικέ ουσίες που ήδη έχουμε απαγορεύσει ή που έχουμε περιορίσει την εμπορία τους ε, προ χώρε, ε, μόνο και μόνο επειδή δεν μπορούν να τι αρνηθούν αυτές οι τρίτες χώρες. Αυτό εννοείται. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να φανταστούμε και να προκαταλάβουμε γιατί απαντούν και όχι κάποιες χώρες αλλά λάβαμε ως απάντηση, για παράδειγμα, ότι υπάρχουν ε, διοικητικές δυσκολίες ε, αλλά βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου πρέπει να αποφασίσουμε αν θα εξαγάγουμε τα πρότυπά μας σε τρίτες χώρες ή αν κατά πόσο θα αποφασίσουν τρίτες χώρες οι ίδιες για το επίπεδο της προστασίας. Εδώ η νομοθεσία για την συνέχιση μετά από ενημέρωση προβλέπει ότι ουσιαστικά η χώρα, η τρίτη χώρα θα πρέπει να αποφασίσει πώς θα ρυθμίσει την αγορά για τα χημικά. Και νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να μείνουμε. Επίσης, νομίζω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε την νομοθεσία όχι μόνο ως ένα κανονισμό, αλλά ως ένα μέσο να ενισχυθεί η διαδικασία αυτή σε τρίτες ε, χώρες, ενώ ελπίζουμε ότι μέσω των προσπαθειών μας, ε, μέσω της ενθήκη, θα ενισχύσουμε τους διαφορούς τομείς προκειμένου να δώσουμε πιο πολύ ουσία στην ε, σύμβαση αυτή. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Καταλαβαίνω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει πολλά καλά πράγματα στον τομέα αυτό και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι κάπως περίεργο το γεγονός ότι ενδεχομένω τώρα να κινούμαστε προ τη λάθος κατεύθυνση. Να θυμόμαστε όμως γιατί πράγμα μιλάμε. Δεν λέμε όπως νομίζω ότι ανέφεραν και κάποιοι προηγούμενοι ομιλητές εμέσως, ότι θέλουμε οι Ευρωπαίοι παραγωγή και εξαγωγής να βρεθούν σε δυσχερή θέση σε σχέση με άλλους. Αυτό που λέμε είναι ότι δεν μπορούν να εξαγάγουν κάτι το οποίο έχει ήδη απογορευτεί εδώ. Πολύ απλά επειδή το κάνουν και άλλοι. Μόνο εφόσον το αποδείξουν ότι υπάρχει έγκριση σε άλλες χώρες. Μπορεί να γίνει για κάποιες χημικές ουσίες, αυτό θέλω να το τονίσω, αλλά δεν μπορούμε να επιτρέψουμε κάτι τέτοιο μόνο και μόνο επειδή έχει συμβεί και στα παρελθόν από άλλους. Νομίζω ότι θα πρέπει επίσης να έχουμε υπόψη μας ποιος είναι ο βασικός ε, σκοπός της σύμβασης του Ροτρεντάμ να προστατεύσει την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Και πραγματικά θα πρέπει να ενισχυθούν οι πτυχέ αυτές και να ακολουθήσουμε αυτό το στόχο. Ευχαριστώ πολύ τους και όδες εισηγητές για την υποστηρίξή σας. Στη γνωμοδότησή μου, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα πιο τεχνικά θέματα και το θέμα της ΕΚΑ, θα πρέπει να βρούμε μία σχετική διατύπωση για την συνεχίση μετά από ενημέρωση. Δεν έχω εγκαταλείψει την αρχική μου γενική θέση, η οποία είναι ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε τον κανονισμό και να καταστήσουμε πιο δύσκολη την χορήγηση μιας τέτοιας απόκλησης. Ευχαριστούμε πολύ, Ντάνιελ, για τις προσπάθειες και για τη δέσμευσή σου για το σημαντικό αυτό θέμα και προθεσμία για τις τροπολογίες 15 Νοεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. Ωραία, λοιπόν. Αγαπητοί συνάδελφοι, Είμαστε και στην ώρα μας και χαίρομαι ιδιαίτερα που έχουμε εδώ την Επίτροπο για την Προστασία του Κλίματος, την Κόνη Χεντεγκάρτ. Σας καλώς ορίζουμε και εσάς και την ομάδα σας. Αυτό έχουμε μόνο κάποιες εβδομάδες πριν από την επόμενη ε, σύνοδο για το κλίμα του ΟΗΕ και έχουμε μπροστά μας και την παρουσίαση του προγράμματος εργασίας ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε κάποιες εβδομάδες θα τεθεί σε εφαρμογή η νομοθεσία για την ανταλλαγή ρήπων στις αερομεταφορές. Έχουμε λοιπόν πολλά ενδιαφέροντα θέματα τα οποία θα ενδιαφέρουν σίγουρα τα μέλη της Επιτροπής μας. Καταρχάς ε, να πούμε ότι ελήφθη σε μια πολύ σημαντική αξιοσημείωτη απόφαση στην Ουάσιγκτον Η απόρριψη της Ευρωπαϊκής Δημοθεσίας από ένα θεσμικό όργανο της ε, Ουάσιγκτον θεωρώ ότι καταδεικνύει άγνοια αλλά και αλαζονία. Αλαζονία γιατί περιμένουμε να εφαρμόζονται τα πρότυπά μας όταν εφαρμόζουμε τα πρότυπα τα ξένα εδώ και άγνοια επίσης αλλά διαπίστωσα ότι υπήρξαν ανακοινώσει τύπου, επιστολές από συναδέλφους, από άλλους κλάδους, οι οποίοι επίσης θέλουν να θέσουν αμφιβόλο την εμπορία ρήπων στις αερομεταφορές. Νομίζω ότι εδώ στην Επιτροπή θα πρέπει να υποστηρίξουμε τι αποφάσει που λάβουμε πριν από κάποια χρόνια και φυσικά θέλουμε να ακούσουμε και τη δική σα θέση. Καλώ ορίσατε λοιπόν κυρία Επίτροπε. Σας δίνω το λόγο. Σας ευχαριστώ. Γιολάινεν, ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για που με προσκαλέσατε για αυτό το διαρθρωμένο διάλογο και ο Πρόεδρος κατά κάποιο τρόπο διευκρίνησε ότι θα ήθελα να ασχοληθώ όχι μόνο με τη διάσκεψη του Δουβλίνου αλλά και με το πρόγραμμα εργασίας και κάποια σχόλια για την ε, αεροπορία και για την ανταλλαγή δικαιωμάτων ε, ρήπων. Έχουμε λάβει πάρα πολλά χρήσιμα σχόλια από την Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος εργασίας ε, για το 2011 και τις προσδοκίες σας ε, για το 2012. Την επόμενη Τρίτη θα υιοθετηθεί το πρόγραμμα εργασίας για το 2012 και ο πρόεδρος Μπαρόζο ήδη στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης ήταν μάλλον σαφής. Ε, είπε γιατί η καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών συνεχίζει να είναι σημαντική. Φυσικά είναι μία από τις βασικές προτεραιότητες μας ακόμη. Σε αυτή την ομιλία αναφέρθηκε ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στην καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες και των πρασίνων τεχνολογιών για να δημιουργηθούν νέε θέσει εργασία. Ε, θα πρέπει ε, οι πράσινοι στόχοι και οι αναπτυξιακοί στόχοι να συμβαδίζουν. Ε, σε μια γραπτή επιστολή μετά από αυτή την ομιλία, σε μια επιστολή που έστειλε ο πρόεδρο Μπαρόζο προ τον πρόεδρο Μπούζεκ, διευκρίνησε ότι ε, και εμεί θεωρούμε ότι οι διαπραγματεύσει για τον προπολογισμό έχουν κέριο ρόλο για να ικανοποιήσουμε αυτέ τι φιλοδοξίε που έχουμε στον τομέα τη προστασία ε, του περιβάλλοντο. Λοιπόν, η πολιτική μα ε, σχετικά με τι κλιματικέ αλλαγέ υιοθετήθηκε όπω και ο δικό χάρη το 2015 προ οικονομίε χαμηλού άνθρακα, καθώ και η ενσωμάτωση του περιβάλλοντο σε όλου του τομεί του προπολογισμού. Για τον οδικό χάρτη τώρα το έχουμε ξανασυζητήσει, δεν θα μπω σε λεπτομέρειε, δεν θα επιμείνω. Παρακολουθήσαμε τι συζητήσει για την προετοιμασία της έκθεσης του Chris Davis και περιμένουμε με ανυπομονησία την συνεισφορά του Κοινοβουλίου. Ελπίζουμε ότι με σαφήνεια υιοθετήσετε την προσέγγιση μας, η οποία όπως ξέρετε έγκυται στο εξή. Χωρίς να έχουμε πολυάριθμες επίσημες συζητήσεις, πώς θα βελτιστοποιήσουμε την ε, δράση μας για την ενεργειακή αποτελεσματικότητα στο μέτρο που αυτό συνιστά ήδη στόχο για την Ευρώπη 2020, για την, στην ανακοίνωσή της για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενισχύσει σημαντικά την ενσωμάτωση των κλιματικών στόχων μέσα σε όλου του τομεί του προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τουλάχιστον το 20% όλου του προπολογισμού θα πρέπει να είναι ανιχνεύσιμο, δηλαδή να αποδεικνύεται σε ποιο βαθμό προωθεί την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων. Ε, έτσι περνάει η Επιτροπή ένα χειρό μήνυμα ότι θα πρέπει να ε, εκπληρούνται οι στόχοι της πολιτικής Ευρώπη 2020 και συγκεκριμένα αυτός ο στόχο για τη μετάβαση προς τις οικονομίες χαμηλή κατανάλωση άνθρακα σχετικά με τα διαρθρωτικά ταμεία, τη γεωργία, την μεταρρύθμιση κοινή γεωργική πολιτική και την υποδομή. Ε, νομίζω ότι φαίνονται με σαφήνεια οι προτεραιότητες ε, της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής. σχεδόν διπλασιάσαμε τα κονδύλια για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή αποτελεσματική στη μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής. Με σαφήνεια φαίνεται ότι προωθούμε την πράσινη συνιστόση. Επίσης βλέπουμε τις αλλαγές στην υποδομή, στην πρόταση για τις υποδομές διότι αποδίδεται ιδιαίτερη έμφαση στις, ε, στους λιμένες, στις χερσαίες μεταφορές, πλωτές μεταφορές κτλ. Δηλαδή δεν υποστηρίζουμε μόνο νέους, πολλούς και νέους αυτοκινητοδρόμους, ε, αλλά εμένουμε στα μέσα μαζικής μεταφορές και στις δημόσιες μεταφορές. Επίσης, ε, εκ παραλλήλου, Προ τα κράτη-μέλη και προ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποστήλαμε την πρότασή μα σχετικά με την οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων, σχετικά με μια μεθοδολογία για τα ορυκτά καύσιμα ε, βάσει τη λογική των αερίων του θερμοκηπίου. Ε, Σα ενδιαφέρει το ζήτημα και φαντάζομαι ότι είδατε πω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ε, με συνοχή αντιμετωπίσει όλες τις οσίες ε, ε, που καλύπτοντας ακόμη και το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο από σχιστόλιθο, ορίζοντας οριακές τιμές για όλες αυτές. Φυσικά θα λάβει η Επιτροπή σας τη συγκεκριμένη πρόταση προς εξέταση μόλις ολοκληρωθούν οι λεπτομέρειες για την οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων. Οι υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής ολοκληρώνουν τώρα την εξέταση σχετικά με την αλλαγή των βιοκαυσίμων, την ε, χρήση σε περίκλειστες ε, χώρες. Ε, εργαζόμαστε άοκνα για να επιτύχουμε ο πρόεδρος ζητά να, από την ομιλήτρια να επιβραδύνει λίγο γιατί δεν μπορούν οι διερμηνείς να την παρακολουθήσουν. Ε, σχετικά με τις αλλαγές στη χρήση της γης ε, συνεχίζουμε τις εργασίες μας ε, και πιστεύουμε ότι μέχρι το τέλος του τρέχοντος θα έχουμε μια νέα πρόταση. Θα ήθελα επίσης θα να σχολιάσω την κατάσταση ως προς την αεροπορία και την περίληψή της στο σύστημα ανταλλαγής δικαιωμάτων λοιπόν, το ETS. Την περασμένη εβδομάδα τα κράτη-μέλη υιοθέτησαν μια μη δεσμευτική και το τονίζω δήληση, παρακινώντας την Ένωση και τα κράτη-μέλη να απόσχουν από την συμπερίληψη των μη ευρωπαϊκών αεροπορικών γραμμών στο σύστημα ETS. Αυτό μπορεί να ξαφνιάζει ορισμένους, αλλά δεν, δεν είναι και κάτι καινούριο, διότι για τις κλιματικές αλλαγές η ΚΑΟ μπόρεσε να συμφωνήσει... Δεν μπόρεσε να συμφωνήσει για πάρα πολλά πράγματα. Συνέχισαν οι συζητήσεις ε, και πιο πολλοί συζητήσει στρέφονταν γύρω από το ότι δεν θέλουν τα κράτη-μέλη και όχι τι θέλουν να κάνουν σε σχέση με αυτό ε, το καύσιμο. Θα ήθελα επίση να σα υπενθυμίσω ότι η επιχειρηματολογία ε, των αντιπάλων μας σε εισαγωγικά ήταν γνωστή τη πάση και συζητήσαμε αυτό το θέμα ήδη όταν η Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν με πολύ μεγάλες πλειοψηφίες ε, το συγκεκριμένο νομοθέτημα. Λοιπόν, η αντίσταση τώρα ε, προβάλλεται από τις ε, ΗΠΑ σε μεγάλο βαθμό και από άλλες τρίτες χώρες και αυτό έχει αρχίσει από το 2005. Γι' αυτό σας είπα δεν είναι κάτι καινούργιο, απλώς πλησιάζει η προθεσμία και κάνουν μια τελευταία προσπάθεια, μπας και τα καταφέρουν. Πάντως, ε, σε μεγάλο βαθμό υπάρχει ε, το λόμπινγκ, πίεση και κινητοποιούνται οι Υπουργοί Συγκοινωνιών, οι Υπουργοί Μεταφορών σε όλα τα κράτη-μέλη λόγω αυτής της πίεσης. Πλην όμως η επιχειρηματολογία είναι ασθενής, διότι ως προς την νομιμότητα των επιχειρημάτων έχουμε τη γνωμοδότηση του 2006 των εξαρτήνων πυρογνωμών, όπου με σαφήνει αναφέρεται ότι όχι, δεν αληθεύει ότι το νομοθέτημά μας, αντιβαίνει στη Σύμβαση Σικάγκο, όχι, δεν αληθεύει ότι δεν θα συνάδει με το UFCC, ε, με την σύμβαση του ΟΗΕ. Όχι, δεν αληθεύει ότι αντιβαίνει στις διατάξει της ΙΚΑΟ. Δεν ευσταθεί ότι πρόκειται για εξοεδαφη, περίπτωση εξοεδαφικότητας ε, και δεν αληθεύει ότι ε, θα μας βοηθήσει από φορολογική πλευράς. Λοιπόν, η προκατακτική γνωμοδότηση σαφέστατα υποστήριζε την αρχική θέση ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης να γνωρίζουμε τώρα που βλέπουμε αυτή την αντίσταση της ΙΚΑΟ να έχουμε επίγνωση του εξή. Οι, οι εμπειρογνώμονες μάλλον ε, της ΙΚΑΟ είχαν καταλήξει σε συναφή συμπεράσματα το 2005. Τώρα δεν αναφέρονται σε αυτά, όμως αληθεύει ότι ήδη το 2004 είχε πει η ΙΚΑΟ το εξή. Καλό θα ήταν να είχαμε αυτό το σύστημα ETS, ε, ανταλλαγή δικαιωμάτων ρήπων δηλαδή, γιατί αυτό το σύστημα είναι πολύ καλύτερο σε σχέση με τα άλλα διαθέσιμα και αν αρχίσετε τώρα θα ήταν λογικό να αρχίσει η λειτουργία του σε περιφερειακό επίπεδο. Τώρα όμως δεν αναφέρονται σε αυτό και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι δεν πρόκειται για άσχετες και ασύνδετες ιδέες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όλα αυτά που προβάλλουμε τώρα είναι διατάξεις της ε, νομοθεσίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Συμβούλιο των Υπουργών Περιβάλλοντος τα ίδια είπα γιατί ε, και τώρα με προσκάλεσε στο επόμενο για να εξηγήσω τη θέση μας. Επίσης, την περασμένη εβδομάδα ε, στο, στην ΙΚΑΟ τα κράτη-μέλη υπεραμήθηκαν τις γραμμή της Ένωσης ε, με ιδιαίτερη πυγμή, δηλαδή δεν αποκλίνει κανείς από την κοινή ε, θέση. Κάτι μας χαροποιεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση φυσικά θέλει να συνεχίσει να ούτως ώστε να καταλήξει σε παγκοσμίω αποδεκτέ λύσεις. Όμως ε, θα σας πω με πάσα ειλικρίνεια ότι την περασμένη εβδομάδα και τις περασμένες μάλλον εβδομάδες και σε ολόκληρη αυτή τη συζήτηση τίποτα καινούριο δεν άκουσα από κανέναν που να αυξάνει τις πιθανότητες μας να βρούμε μια παγκόσμια λύση για τις κλιματικές αλλαγέ σύντομα. Εμείς πάντως δεν αποτελούμε εμπόδιο για την εξέβρεση λύσης. Τώρα για τι βασικέ ε, προτεραιότητε στρατηγική 2020. πρώτον έγκαιρη ε, εφαρμογή του ενεργειακού και κλιματικού πακέτου. Αυτό θα συνεχίσει να αποτελεί προτεραιότητα κυρίω εν ώψη τη τρίτη ε, φάσης του ETS που θα αρχίσει το 2013. Δεύτερον, προετοιμάζουμε πολυάριθμε πρωτοβουλίε στον τομέα τη κλιματική δράση σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση, Θα αναθεωρήσουμε τον κανονισμό για τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά και το διοξίδιο του άνθρακα είναι σημαντικά αυτά τα νομοθετήματα για να μειωθούν οι εκπομπέ ε, ε, κατά τι μεταφορέ ε, και για να έχουμε μεγαλύτερη κοινοτομία στον τομέα. Σχετικά με τι εκπομπέ τι θαλάσσιε μεταφορέ, αφέστατα τα προτιμούμε την παγκόσμια σε κλίμακα σε δράση και τώρα εκινούμε τι δράσει μα για να καταθέσουμε εμεί πρόταση αν μέχρι το τέλο του 2010 δεν έχει εγκριθεί διεθνή συμφωνία που να συνάδει πλήρω με αυτά που μα είχε ζητήσει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μόλι άκουσα τώρα από την τρίτη συνεδρίαση του πάνελ των εμπλεκόμενων φορέων όπου συζητούμε δηλαδή με όλους τους εταίρους ε, για την άγουσα που θα ακολουθήσουμε ε, συνειδητοποιούμε ότι σημειώνονται εξελίξεις. Ε, επίσης, ο κανονισμός για το φυσικό αέριο, όπου ε, ο στόχος μας ε, είναι αποτελεσματική ε, μείωση των εκπομπών με καλή σχέση κόστους ωφέλους. Επίσης θα προετοιμάσουμε την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προσαρμογή που προβλέπεται για το 2013. Οι Ιταλοί, Γάλλοι και άλλοι συνάδελφοι υπό το φως ε, των εξελίξεων στις χώρες τους νομίζω θα περιμένουν με ανεπομονησία τι εξελίξει. Τέλος, αλεξίου σημαντικό, επίσης για το 2012 θα πρέπει να συνεχίσουμε δραστήρια να εμπλεκόμαστε στις διεθνείς προματεύσεις για την επίτευξη στόχου σχετικά με μια νομικά δεσμευτική συμφωνία ε, ε, και ελπίζω ότι θα καταλήξουμε σε κάτι πριν από τον Τέρμπεν θα ήθελα να σχολιάσω αυτή τη διάσκεψη στον Τέρμπαν για τις κλιματικές αλλαγές ε, λίγο περισσότερο. Νομίζω ότι είναι δίκιο να πούμε ότι η θεώρησή μας, ε, η θεώρησή μου ε, συμβαδίζει ε, με τα επιμέρους στοιχεία της νομοδότησης του Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ που εργαστήκατε σκληρά και υιοθετήσατε αυτή την πρόταση ψηφίσματος που από ό,τι κατάλαβα θα ψηφιστεί την επόμενη Τρίτη στην Ολομέλεια στο Στρασβούργο. Λοιπόν, το Ντέρμπαν είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να προοδεύσουμε, να βασιστούμε στην σύμβαση της Κανκούν ήμουν ε, και στα αποτελέσματα της διάσκεψης της Κομπενχάγης από πέρσι. Ξέρουμε όλοι ότι δεν θα είναι ε, το τέλος του δρόμου μας, αν θέλετε, εδώ Ντέρμπαν. Ε, θα συγκεκριμενοποιήσουμε τη συμφωνία της Κανκούν και θα πραγματευτούμε τα εκρεμή, τα ζητήματα που παρέμειναν εκρεμή μετά την Κανκούν. Ένα από αυτά είναι το θέμα της νομικής μορφής. αυτό πάλι θα τεθεί επιτάπητος η Ευρωπαϊκή Ένωση Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να υπάρχει ένα ε, συνεκτικό, πλήρες ε, πλαίσιο, νομικό, νομικά δεσμευτικό πλαίσιο που θα λειτουργεί σε δύο βαθμούς. Φυσικά θέλουμε να γίνεται σεβαστό το πολυμερές πλήσιο που είχε προβλεφθεί από το πρωτόκολλο του Κιώτο όμως. Η δεύτερη περίοδος ανάληψη υποχρεώσεων, η δεύτερη φάση δεν ε, πρόκειται να περιορίσει την αύξηση στους δύο βαθμούς ε, για την υπερθέρμανση του πλανήτη. Ακόμη και η Νορβηγία και η Ελβετία ε, θα μπορούσαν να εισέλθουν σε αυτή τη δεύτερη περίοδο εφαρμογής, αλλά αυτό δεν λύνει το πρόβλημα. Τι θα γίνει με αυτά τα 80 κάτι της με ποιο με τι θα γίνει με τι υπόλοιπε χώρε, ε, πώ θα αναλάβουν τι αντίστοιχε δεσμεύσει. Το θέμα δεν είναι επιλέξουμε αν θα ακολουθήσουμε το Κιώτο ή όχι. Το διακύβευμα του Ντέρμπαν ναι, είναι ακριβώ να υπερβούμε το πρωτόκολλο του Κιώτο και αυτό το χάσμα που δημιούργησε, ούτω ώστε όλε οι χώρε, ε, και οι αναπτυσσόμενε ε, και οι ανεπτυγμένε, να αφοσιωθούν στην επίτευξη των στόχων που θα έχουν αναλάβει σε αυτό το παγκόσμιο πλαίσιο. Και άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση προτίθεται να εξετάσει μια δεύτερη περίοδο αλλά στα πλαίσια ενός ε, γενικότερου πακέτου, γενικότερου ε, πλαισίου. Ε, και προϋποθέτει αυτό αναβάθμιση των κανόνων του Κιώτο, και συγκεκριμενοποίηση των κανόνων που προβλέπονταν εκεί πέρα, των κανόνων EFSA. Ε, για το νομίζω ότι χρειαζόμαστε σαφή οδηγικό χάρτη, ε, σαφέστατο χρονοδιάγραμμα, ούτω ώστε είπαμε να είναι περιεκτική, διεξοδική, πλήρη ε, η συμφωνία, να είναι πακέτο, να είναι νομική, νομικά δεσμευτική και να βασίζεται στην αρχιτεκτονική του Κιώτα και να εμπλουτιστεί από κανόνε για του οποίου θα συμφωνήσουμε στο Ντέρμπαν. Αυτή τη στιγμή με του εταίρου μα και με τι αναπτυγμένε και με τι αναπτυσσόμενε χώρε με αυτό ασχολούμαστε. Με ποια βήματα θα προτείνετε να κάνουν προ αυτή την κατεύθυνση για να προαγάγουν μια κοινή και φιλόδοξη λύση. Πριν σταματήσω θα ήθελα ε, να σας πω ότι πιστεύω πως ε, τους τελευταίους ε, μήνες υπήρξαν κάποιες εξελίξεις προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή να υπάρξει μεγαλύτερη κατανόηση, αν θέλετε, για θέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο συγκεκριμένα, πολλές αναπτυσσόμενες χώρες κατανοούν ότι εάν αναλάβουμε εμεί τη δεύτερη περίοδο ανάληψη υποχρεώσεων άνευ όρων, το πρώτο που θα συμβεί είναι ότι η πίεση δεν θα βαραίνει πλέον τους ώμους ε, των βασικών, ε, των μεγαλύτερων οικονομιών, είτε πρόκειται για ανεπτυγμένες, είτε πρόκειται για αναπτυσσόμενες χώρες. Οπότε ε, η δική μας δουλειά είναι να πετύχουμε τη σωστή συμφωνία φυσικά ε, αυτός ο δικός ε, χάρτης ε, δεν σημαίνει ότι θα τα αφήσουμε όλα ανοιχτά. Γι' αυτό σας μίλησα για το χρονοδιάγραμμα. Θα πρέπει να θέσουμε κάποια όρια, αλλά... Αυτό είναι ένα από τα βασικά ζητήματα του Ντέρμπαν και νομίζω ότι επ' αυτού την χάνει μεγαλύτερε αποδοχή η θέση τη Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το COP15. Οι περισσότεροι εταίροι καταλαβαίνουν γιατί είναι λογική η πρότασή μα, αλλά ε, διότι συγγνώμη, συνειδητοποιούν τη συνεισφορά αυτού του σχεδίου για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Άλλο κέριο σημείο είναι παρακολούθηση τη σειρά αποφάσεων που λήφθησαν στο Κανκούν για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό συμπεριλαμβάνει κέρια σημεία, παραδείγματο χάρη μετανάστευση, ε, ελαχιστοποίηση, mitigation. Επίση, ε, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα τη ανάληψη υποχρεώσεων για τι παγκόσμιε εκπομπέ και αύξηση τη φιλοδοξία, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνουμε του κανόνε σε Κανκούνε για καλύτερα αποτελέσματα στην καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Άλλο θέμα είναι η χρηματοδότηση. Προφανέστατα εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή και τα 27 κράτη-μέλη να ικανοποιήσουμε τις υποχρεώσεις ε, που αναλάβαμε στην Κοπενχάγη. Ε, καταλαβαίνετε ότι αυτό επηρεάζει το κλίμα όλων των διαπραγματεύσεων και γι' αυτό φέτος ε, όπως και πέρσι ε, θα αναφέρουμε λεπτομερώς τι υποστηρίζουμε για το 2011, πόσα κονδύλια έχουμε, με ποιο τρόπο μπορούμε να καλύψουμε τις υποχρεώσεις μας Κοπενχάγης, πόσα χρησιμοποιούνται για την προσαρμογή, πόσα για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών, πόσα για τη δασοκομεία, για να ε, γνωρίζουμε ότι πώς οι αναπτυσσόμενες χώρες, οι πιο ασθενείς χώρες θα μπορούσαν να δεχτούν την πρότασή μας για να καταφέρουμε να βρούμε μια ισορροπία. Αυτό το κομμάτι ε, της χρηματοδότησης είναι σημαντικό γιατί στον Τέρμπαν ε, θα ε, πρέπει να βρούμε πώς ακριβώ θα βρούμε τα 100 δίσε δολάρια ετησίως μέχρι το 2020 από ε, δημόσιες, ιδιωτικές και καινοτόμες πηγές χρηματοδότησης. Όμως υπάρχει και το θέμα είναι εντάξει για τα κονδύλια, εντάξει για την περίοδο μέχρι το 2020 και τι θα γίνει στην περίοδο ανάμεσα στο 2013 και το 2020 για να καλύψουμε αυτή την περίοδο προετοιμάζουμε εδώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου ένα συγκεκριμένο κομμάτι για το EES Και νομίζω ότι με αυτέ τι δράσει μα έχουν καταλάβει οι εταίροι ότι θα παράσχουμε χρηματοδότηση για αυτή την επταετή περίοδο, το 2013 μέχρι το 2020 δηλαδή. όμω, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι δεν περιμένουμε από τον Τέρμαν μόνο να τηρήσει τι ε, υποχρεώσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση ω προ τη χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση θα πρέπει να είναι ένα κομμάτι ενό συνολικού πακέτου. Δηλαδή, όταν έχουμε όταν λαμβάνουμε ε, δεσμεύσεις ε, δεν μιλάμε μόνο για τη χρηματοδότηση. Επίση πρέπει να μεριμνήσουμε ότι τα κονδύλια ε, χρησιμοποιούνται για συγκεκριμένου στόχου σε συγκεκριμένες χώρες και γι' αυτό σα είπα ότι θα πρέπει να δεχτούμε, να καλύψουμε τι δεσμεύσει για τη χρηματοδότηση στα πλαίσια ενό συνολικού πακέτου. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε Επίτροπε Χέντιγκάρτε. Για την δέσμευσή σα, για την μεγάλη σα αυτή απασχόληση με το μεγάλο αυτό θέμα και θα πρέπει να πω ότι υποστηρίζω πλήρως τι απόψει σα για το σύστημα εμπορίας ρήπων και τις μεταφορές. Τα επιχειρήματα κατά τη συμπερίληψη δεν είναι καινούρια και τα λόμπι πάντα επαναλαμβάνει τα ίδια επιχειρήματα. Προσπαθεί τελευταία στιγμή να παρακολύσει την νομοθεσία. Και τελικά όταν θα εφαρμοστεί θα δούμε ότι δεν θα είναι τόσο κακό όσο υποστηρίζουν οι πολέμοι του συστήματος. Ωραία λοιπόν για το το 2 ναι ή όχι. Νομίζω ότι η συζήτηση αυτή θα συνεχιστεί. Και τώρα, συνάδελφοι, έχουμε 11 μέλη της Επιτροπής μας που θέλουν να πάρουν το λόγο. Δύο λεπτά για τον καθέναν. Σας παρακαλώ να σεβαστείτε το χρονικό όριο για να μιλήσουν όλοι. Να ξεκινήσουμε και πάλι με τους συντονιστές. Δύο λεπτά ο καθένας. Ευχαριστώ κύριε Ζέμπερ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και την Κόνη Χέντεγκαρ για την παρουσίασή σας. Μια συγκεκριμένη ερώτηση Διαβάσαμε σήμερα στην Financial Times ότι για τον οδικό χάρτη το μοντέλο που χρησιμοποιείται είναι πανεπιστημιακό μοντέλο και ότι δεν είναι κάτι το οποίο πραγματικά μπορεί να εφαρμοστεί. Θα μπορούσατε πραγματικά να μου διευκρινίσετε κυρία Επίτροπε τι γίνεται. Γιατί για τόσα σοβαρά ζητήματα για το 2050 θέλουμε να διαθέτουμε διαφανή μοντέλα και μάλιστα με αξιοπιστία. Κατά δεύτερον, συμφωνώ με την εκτίμησή σας ότι αφορά το Κιώτο. Το θέμα δεν είναι μόνο να συνεχίσουμε την χρηματοδότηση ως Ευρωπαίοι και μόνο. Όχι, θα πρέπει να συμφωνήσουμε επί ενός συνολικού πακέτου και αυτό αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία τα οποία θα κληθούμε να διευκρινίσουμε στο Τέρμπαν. Να συγχαρώ επίσης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το mainstreaming σε ό,τι αφορά τα τα ταμεία και τα ΚΑΠ, νομίζω ότι συνολικά θα πρέπει σε ευρωπαϊκό επίπεδο να προσπαθήσουμε να θέσουμε στόχους. Γίνεται συζήτηση για την οδηγία, για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Θέλουμε λοιπόν δεσμευτικούς στόχους, αλλά όσο πιο πολύ ευελιξία γίνεται για τα κράτη-μέλη, γιατί θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι διαφορές που υπάρχουν και ελπίζω πραγματικά τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να συμμετάσχουν σε ό,τι αφορά θέματα χρηματοδότησης τώρα. Είμαι ρεαλιστής ε, και απεσιόδοξος. Κοιτώντας τι γίνεται τους τελευταίους ε, μήνες, τα τελευταία χρόνια, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, ελπίζω να τα έχουμε υπερπηδήσει σύντομα. Η Μέρκελ λέει σε 10 χρόνια ο Φιγιόν από τη Γαλλία λέει ότι βρισκόμαστε στο σημείο καμπής. Θα πρέπει να τα έχουμε όλα αυτά υπόψη τα θέματα χρηματοδότησης. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Η Λίντα Μακέβαν διακόπτει ο Πρόεδρος γιατί δεν έχουμε χρόνο. Λυπάμαι, λυπάμαι πολύ. Ευχαριστώ που επιμένετε σε θέματα αερομεταφορών γιατί Ξέρετε, σας υποστηρίζουμε σχεδόν όλοι εδώ και σε θέματα σχιστόλιθων. Και το θέμα που έθεσε ο κύριος Ζέμπερ αναφέρθηκε υποστήριξη προς τον Καναδά στην εφημερίδα. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Και για τη βιομάζα να σας ρωτήσω. Δεν θέλουμε να δημιουργηθεί παρόμοιο χάος ό,τι αφορά την βιομάζα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τέλος του χρόνου θα παρουσιάσει κάποια κριτήρια βιωσιμότητας. Ε, τα πιο πολλά κράτη-μέλη δεν έχουν ε, ε, ουσιαστικά παραγωγή βιομάζας, αλλά υπάρχει εισαγωγή βιομάζας, χωρίς να ξέρουμε κατά πόσο είναι βιώσιμη η παραγωγή της, από πού προέρχεται, θα υπάρχουν λοιπόν σχέδια βιωσιμότητας για τη βιομάζα στην Ευρώπη. Ευχαριστώ κυρία, ο κύριος Κράμερ. Ευχαριστώ πολύ σύντομα για το θέμα της ε, αερομεταφοράς και της συμπερίληψης στο ETS. Θα ήθελα να τονίσω ότι δεν ήταν κάποιο θεσμικό όργανο στην ε, Ουάσιγκτον. Όχι, ήταν οι κυβερνήσεις όλου του κόσμου που είναι υπεύθυνοι για τις αερομεταφορές. Αυτές έλαβαν την απόφαση. Καταρχάς δεν είναι δεσμευτικό το ψήφισμα, αλλά αποτελεί ένα χειρό μήνυμα παρόλα αυτά. Και δεν θα πρέπει να μας εκπλήσει ότι ελήφθη αυτή η απόφαση μετά το προηγούμενο Σαββατοκυριακό. Θα ήθελα να ρωτήσω μήπως ε, μετά την απόφαση του ΙΚΑΟ θα πρέπει να υπολογίσουμε ότι τα κράτη-μέλη που έχουν εκφράσει αντιθέσεις θα εμείνουν στις αντιθέσεις και ότι δεν πρόκειται να υπάρχει καμία πρόταση για σχετικά μέτρα. Υπάρχουν καν τρίτα μέλη που έχουν κάνει, τρίτα κράτη που έχουν κάνει προτάσεις για αντίστοιχα μέσα και μήπως ε, πολιτικά αυτό είναι επιζήμιο, μήπως θα πρέπει να διαπιστώσουμε μετά τις εξελίξεις των τελευταίων μηνών ότι η προβληματική των τρίτων κρατών ήταν κάτι που υποτιμήσαμε σημαντικά. Φτάνει να επιμείνουμε και να σκεφτόμαστε ας άσπρο στο θέμα αυτό. Μήπως αυτό διπλωματικά και οικονομικά βλάπτει την Ευρώπη. Ε, ευχαριστώ, Καρλ Σλούτερ. Ναι, σας ευχαριστώ. Χαίρομαι που το έχετε πάρει κατάκαρδα το θέμα της ε, αεροπορίας. Ε. Υπάρχει το πρόβλημα επίσης με τους στόχους του 2013 για τις θαλάσσιες μεταφορές. Θα πρέπει να δείξουμε στον υπόλοιπο κόσμο ότι ούτως ή άλλως θα τα αναλάβουμε αυτά τα μέτρα για να τους εμπνεύσουμε. Για το Λουσιεφ, Θεωρείτε ότι μπορεί κάποιοι να χρησιμοποιήσουν ως πρόσχημα τη δασοκομεία για να ξεφύγουν από το ETS και από τους εθνικούς στόχους για την ανταλλαγή ρήπων. Ε, τώρα για την ασφαλτούχο άμμο, για τις ε, γεωτρήσεις σε ανοιχτή θάλασσα, για το αέριο από το σχιστόλιθο και όλα αυτά τα θέματα. Φοβάμαι ότι ε, θα τραβήξουν πάρα πολλοί διαπραγματεύσεις. Ε, κατά τη γνώμη σας, ε, μια φιλόδοξη πολιτική αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών μπορεί να συνδυαστεί με την χρήση των πόρων για αυτά τα ζητήματα. Δεν το νομίζω. Ε, οι μελέτες ε, δείχνουν ε, έχουμε, ότι έχουμε 2 με 3% να τηρήσουμε αυτό το στόχο των 2 βαθμών. Μέχρι το 2005 θα πρέπει να έχουμε φτάσει σε μηδενικά επίπεδα για τις ε, ε, εκπομπές. Άρα τι μπορούμε να κάνουμε για τις επενδύσεις σε αυτούς τους τομείς, ε, γιατί η απόσβεση προβλέπεται για πολύ αργότερα από την ημερομηνία που προβλέπεται θα σταματήσουν την παραγωγή. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να να, με τη σειρά μου και εγώ να σας ε, συγχαρώ για τη θέση σας, ε, συγκεκριμένα για την ασφαλτούχο άμμο και για το ETS ε, στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας. Δύο παρατηρήσεις έχω να κάνω. Μία για, συγκεκριμένα για το πρωτόκολλο του Κιώτο. Εδώ είμαι. Θα είναι ιδιαίτερα επιζήμιο νομίζω αν δεν εισέλθει σε δεύτερη περίοδο ανάληψη υποχρεώσεων η Ευρωπαϊκή Ένωση εν ώψη του Ντέρμπαν, διότι θα είναι σφαλμένο το μήνυμα που θα περάσουμε στις ε, αναπτυσσόμενες χώρες ε, και ενδέχεται να προκαλέσει μια αρνητική ε, αντίδραση από πλευράς κάποιων που, από τους οποίους περιμένουμε όμως θετικές αντιδράσεις. Μιλήσατε για την ε, μεσαία λύση, την χρυσή, το που θα επιδιώξουμε στον Τέρμπαν. Μιλήσατε για το χρονοδιάγραμμα, για τον ειδικό χάρτη κτλ. Ε, μπορείτε να μου πείτε στις συμφωνίες ε, της, ε, ε, του Κανκούν είχαμε αντίστοιχες, αντίστοιχους στόχους αν θέλετε για χρονοδιαγράμματα και τα λοιπά μας βοήθησαν εν αναμονή του Ντέρμπεν μήπως Μήπως αν περιοριστούμε σε ημίμετρα αυτού του τύπου ε, μήπως αυτό έχει το αντίθετο αποτέλεσμα, μήπως δείξει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν είναι αρκετά σοβαρή ως προς τους στόχους. Ε, είναι αυτό που σας έλεγα και προηγουμένω ότι μπορεί να περάσουμε αρνητικά μηνύματα σε αναπτυσσόμενες χώρες. Ε, και ε, Ξέρετε, όταν ακούσαμε τελευταία παρουσία στην Επιτροπή Περιβάλλοντο, η τελευταία πρόταση ήταν μην, μη πάτε καν στον Τέρμπαν, ούτε δεν αξίζει, δεν πρόκειται να καταφέρετε τίποτα. Ευχαριστώ, Κάρι Φρόντ. Yeah, Äh ναι, Κοιτώντα τα τελευταία συμπεράσματα, την τελευταία ανακοίνωση του Συμβουλίου, δεν είμαι βέβαιο κατά πόσον υπάρχει μια απάντηση για τον Τέρμπαν. Πολλά έμειναν ανοιχτά σε ό,τι αφορά το θέμα του Κανκούν, τη συμφωνία του Κανκούν και το πώ ε, θα προωθήσουμε μια παγκόσμια αγορά για τους ε, τα θέματα αυτά. Δεν είμαι βέβαιο ότι ω Ευρωπαίοι έχουμε δίκιο. Στην Κοπενχάγη ήταν αρκετά αλαζονική η στάση μα. Θα ήθελα να ακούσω πώ είναι δυνατόν στο Κιώτο 2-3, όπω θέλετε επιδετώ, να γίνει μία ε, σύνδεση με τι λιγότερο αναπτυγμένε χώρε. χώρες θα υπάρξει νομική βάση. Θα ήθελα να μάθω με όλες τις καλές προθέσεις που έχουμε, με όλες ε, τις προτάσεις που μπορούμε να κάνουμε, Αλλά ξέρετε, οι προθέσεις δεν αρκούν. Η πρακτική στρατηγική. Ποια είναι για να προωθήσουμε συγκεκριμένα θέματα. Ευχαριστώ, Ματίας Κρότα. Ευχαριστώ, Κόνι Χέντεγκαρτ, και για τη δέσμευσή σας. το γεγονός ότι η Επιτροπή επέμεινε τόσο πολύ σε ό,τι αφορά τις αερομεταφορές στο σύστημα ETS. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ σε μια συγκεκριμένη αναφορά που κάνετε για, την, ε, για τα αυτοκίνητα και για το 2014 σε ό,τι αφορά την εκπομπή του του άνθρακα. Σε όλο το κύκλο ζωής των αυτοκινήτων γιατί αυτό είναι ο στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να δούμε πώ παράγεται ένα αυτοκίνητο και πόσο, ε, μάλλον και πόσο κατά πόσο θα μπορούσαν να κατασκευαστούν αυτοκίνητα χωρίς ε, του άνθρακα. Αυτή η, η οικολογική κοινοτομία την οποία διαπραγματευθήκαμε σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις. Έχουμε προχωρήσει αρκετά στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά την νομοθεσία και την προστασία του κλίματος, αλλά πάντα απογοητευόμαστε στο διεθνές προσκήνιο. Μήπως χρειάζεται μεταξύ των διασκέψεων να ξεκινήσουμε μια διπλωματία για το κλίμα στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, γιατί κάποιες φορές έχω την αίσθηση ότι είσαστε δεσμευμένοι, αγωνίζεστε, αλλά κάπου είναι τόσο ψηλό το τείχος που καλείστε να αντιμετωπίσετε από την άλλη πλευρά, που ίσως θα χρειαζόταν μια κλιματική διπλωματία μεταξύ των συνόδων, προκειμένου να μην αποτελεί μόνο ένα μικρό βήμα επιτυχίας κάθε τέτοια σύνοδος. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και καλώς ήρθε η Επίτροπος εδώ. Με πάρα πολύ προσοχή παρακολούθησα τα όσα μας είπε. Και καταλαβαίνω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κάνει μεγάλη προσπάθεια για να αντιμετωπίσει τα αέρια του θερμοκηπίου και όσον αφορά τις θαλάσσιες μεταφορές, τις εναέρειες, τις ελαφρές μεταφορές κλπ. Προσπάθειες προσπάσα πάσα κατεύθυνση. Θέλω όμως να επανέλθω σε ένα ιδιαίτερο ζήτημα, το οποίο κατά τη γνώμη μου σε τοπικό επίπεδο τουλάχιστον έχει μεγάλες επιπτώσεις επί του κλίματος. Είμαι από τη Βενετία και εκεί υπάρχει ένα σχέδιο για τον άνθρακα. Για 85 ΜΒ μιλάμε για 10 εκατομμύρια τόνους διοξίδιο του άνθρακο που ε, ετησίως παράγονται. Μέσω θαλάσσης θα μεταφέρεται ε, ο άνθρακας από την Ινδονησία. Έτσι λοιπόν αν θέλαμε να συλλέξουμε αυτόν τον άνθρακα θα κόστιζε ένα δισεκατομμύριο. Δεν γίνεται. Πρόσφατα λοιπόν η Ιταλική κυβέρνηση ενέκρινε ένα διάταγμα και η περιφέρεια Αυτό λέει. Της, ε, η περιφέρεια λοιπόν επίσης ενέκρινε κάτι αντίστοιχο. Οι πολίτες τώρα πιστεύουν ότι η μονάδα αυτή δεν πρέπει να χτιστεί γιατί αντιβαίνει στις ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι για τον περιορισμό των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Η Ιταλία πάλι θέλει να αντιμετωπίσει ε, τις επιπτώσεις στο κλίμα είναι συνολικά 2,5 ε, δισεκατομμύρια. Δεν θα ήταν καλύτερα να τα ξοδέψουμε για τι εναλλακτικέ ενέργειε. Πρόεδρο Διακόπτη, καταλάβαμε ε, τι λέτε. Ερώτηση, κύριε Σένε. Λοιπόν, τι θα κάνει η Επιτροπή, θέλετε να ρωτήσει τώρα, κύριο Ασένη. And... Καλώ ορίσατε, Επίτροπε, και σα ευχαριστώ που ήρθατε εδώ πέρα, στην Επιτροπή μα. Σα αποστήλαμε μια επιστολή για την δεύτερη προγραμματική περίοδο, την οποία και υπέγραψαν και άλλα μέλη. Και ελπίζουμε να τύχει μεγαλύτερη ε, υποστήριξη και εκπροσώπηση. Είναι σαφέ ότι δεν έχουμε κάτι να χάσουμε. Δεν, αλλάγουμε, δεν αλλάζουμε πολλά σε ό,τι αφορά τις ε, υποχρεώσεις μας. Και αν χάσουμε την ε, ορμή για μια δεύτερη τέτοια περίοδο δεσμεύσεων, είναι σαφές ότι δεν θα προκύψει νομικός δεσμευτική α, ε, συμφωνία με τις α, ε, αναπτυσσόμενες χώρες. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν ε, γιατί ακολουθούμε την τακτική που ακολουθούμε, γιατί δεν συνεχίζουμε την πίεση, την άσκηση πίεσης. Κάτι άλλο. Ένα από τα θέματα πέρα από την αερομεταφορά Έχουμε δέσμευση. Να εφαρμόσουμε σχετική νομοθεσία μέχρι το 2014. Έγινε μια νέα συμφωνία στην IMO το καλοκαίρι και τουλάχιστον μια κυβερνητική οργάνωση ανέφερε ότι ήταν η πρώτη συμφωνία από ένα βιομηχανικό κλάδο που μπορεί να οδηγήσει σε μείωση μέχρι και 20% μέχρι το 2030. Ο δικός χάρτης μας λέει 40% μέχρι το 2050. Θα ήθελα λοιπόν κάποια πρώτα σχόλια, αν θέλετε να μου κάνετε. Ευχαριστώ, κύριος Λίζα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την κυρία Επιτροπό για τις ε, σαφείς κουβέντες. Τρεις ερωτήσεις, πολύ σύντομα. Σε ό,τι αφορά την ενεργειακή αποδοτικότητα και την πρόταση του Επιτρόπου Oettinger, συζητάμε την πρόταση αυτή στο Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή και συζητάμε κατά πόσον οι απόλυτες μειώσεις ε, που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεπάγονται και κάποιο σχετικό στόχο για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Συμφωνείτε ότι δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο ύφεση και ότι βρισκόμαστε σε επίπεδο 30%, θέλουμε μάλλον επίπεδο 30% μείωση στις εκπομπές, αλλά ίσως ε, τελικά η βιομηχανία καταφέρει μόνο 20% σε ό,τι αφορά την διαρροή άνθρακα στις ε, έμεσες ε, εκπομπές. Θα πρέπει να υπάρξει απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθοριστική προκειμένου σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τη και την βιομηχανία αλουμινίου να υπάρχει και ένα σχέδιο για τις αερομεταφορές τώρα. Υποστηρίζω τις απόψεις σας όπως και πολλοί συνάδελφοι. Να προσθέσω δύο επιχειρήματα. Η επιβάρυνση του ETS για τις διαατλαντικές πτήσεις είναι πολύ περιορισμένη. Δύο ευρώ για παράδειγμα. Συνεπάγεται για μία πτήση από τη Γερμανία. Ενώ ας πούμε άλλα στοιχεία επιβαρύνουν και πολύ περισσότερο τα αεροπορικά εισιτήρια. Είναι ένας εύκολος στόχος. Το ερώτημα του γιατί έχουμε τόσους λίγους συμμάχους. Είπε ο κύριος ε, Μπαρός ότι θα πρέπει να κάνουμε διαφήμιση για την ε, θέση μας αυτή στο Δέρμαν. Η κυρία Χάση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σύμφωνο με τους συναδέλφους που ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, επιδείξει θάρρος σε ό,τι αφορά το σύστημα εμπορίας ρήπων. Και θα ήθελα να εκφράσω και εγώ την υποστήριξή μου σε ό,τι αφορά τη συμπερίληψη του θέματος του κλίματος σε όλο τον προϋπολογισμό της Ένωσης. Αυτό που δεν έχουμε ακόμα ερωτήσει είναι ο σύνδεσμος μεταξύ ενεργειακής αποδοτικότητας και του συστήματος εμπορίας ρήπων. Ξέρουμε ότι αν ο στόχος ε, της ενεργειακής αποδοτικότητας επιτευχθεί, θα έχουμε υπερβολικά δικαιώματα ε, εκπομπής ρήπων στο σύστημα ETS και υπάρχει κίνδυνος να καταρρεύσει το σύστημα. Και σε διάφορα αφορά τις πράσινες επενδύσεις. Ρωτώ λοιπόν αν σκοπεύετε να προσαρμόσετε τα τα όρια του ETS προκειμένου να συνάδει και με την πολιτική βούληση την οποία εξέφρασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά την ε, οδηγία για την ενεργειακή αποδοτικότητα και επίσης να συνάδει με την προσέγγιση αποδοτικότητας κόστους σε ό,τι αφορά τη μείωση των εκπομπών μέχρι το 2050. Ευχαριστώ κύριε Σιωρίτινσον. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θέλω να σας ρωτήσω κύριε Επίτροπε. Τι κριτήρια επιτυχίας βάζετε για τον Τέρμπαν. Είναι σημαντικό να είσαστε συγκεκριμένοι. Ξέρω ότι υπάρχει ένας κίνδυνος. Αν δεν πετύχουμε τότε θα κρυθεί αποτυχία. Αλλά από την άλλη είναι πολύ σημαντικό εμείς να ξέρουμε ότι και η διαδικασία των ΗΠΑ πρέπει να προχωρήσει αλλά και το ότι είναι χρήσιμη. Μετά την Κοπεχάγη Πολλοί είπαν ότι έχει λήξει η διαδικασία, έχει πεθάνει η διαδικασία κόπ. Πολλοί ε, άλλοι είπαν πως όχι. Λοιπόν, στον Τέρμπαν, αν δεν έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα να επιδείξουμε, φοβάμαι ότι η πίεση θα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Και σε σχέση με αυτό, όταν μιλάτε για το θέμα του Κιώτο, εσείς περιμένετε να καταλήξει κάπου στον Τέρμπαν. Δεν είμαι σίγουρος τι ακριβώς προβλέπετε. Μιλάμε για έναν οδικό χάρτη αντί για την δέσμευση ή θα αποτελεί μέρος μια περίοδος ε, δέσμευσης για ε, τον οδικό χάρτη, θα είναι μέρος του. Θέλετε να υπάρχουν υποχρεώσεις και αν είναι υποχρεώσεις ε, γιατί πράγμα θα είναι για το ΠΙΚ, για την ενεργειακή απόδοση, για τι πράγμα μιλάμε. Και τέλος κάτι πιο πρακτικό. Πώς βλέπετε το ρόλο της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εμείς βέβαια είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τις δικές σας προσπάθειες, τον τρόπο που εκφράσετε κτλ. Σύμφωνοι, αλλά δεν είδαμε μεγάλη αλλαγή ε, τώρα με τη νέα συνθήκη δεν θα έπρεπε να προσκληθεί αν μη τι άλλο ο πρόεδρος της Επιτροπής μας στις ονήσεις που γίνονται με το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Πολύ καλή ερώτηση αυτή, λέει ο πρόεδρος. Και τον αντιπρόεδρο, γιατί όχι. Να είναι ανοιχτή πόρτα. Η Μαργαρέτα είναι η τελευταία ομιλήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω δανέζικα. Αγαπητή Κόνη, πρώτα απ' όλα Υποστηρίζω απόλυτα τις δικές σου προσπάθειες. Ξέρω τι έχεις κάνει ε, στον ΙΚΑΟ. Ήταν πραγματικά εξαίρετο αυτό τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας. Τώρα, τα χρήματα αυτά για τα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται. Τι θα δώσει αυτό είναι κάτι μήπως που θα μείνει μόνο στα λόγια, θα είναι υποσχέσεις. Ξέρω επίσης ότι θέλεις να γίνουν τα πράγματα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί αν η κάθε χώρα δεσμευτεί χωριστά, δεν έχουμε την εγγύηση ότι το συνολικό ποσό τελικά θα επιτευχθεί. Υπάρχει πραγματικά μια κοινή στρατηγική σε αυτό το τομέα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ακούστηκαν διάφορες ερωτήσεις όσον αφορά τη στρατηγική μας, τη τακτική μας σχετικά με το Κιώτο 2. Εγώ φαντάζομαι ότι θέλετε περισσότερα ακόμα. Η πρόταση ίσως δεν είναι αρκετά καλή. Πηγαίνουμε μέχρι το 13, 14, δεν μέχρι το 15. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως έχει κάτι να προσφέρει. Γιατί το πακέτο για την ενέργεια και το κλίμα είναι νομοθεσία. Είναι δηλαδή 20% που έχουμε κάνει μονομερός και δεν έχουμε τίποτα να προσφέρουμε. Τι θα τους πούμε, περιμένετε το 2015 και τότε και για τι πράγμα, με τι στόχο. Το ψήφισμά μας που θα ψηφίσουμε την επόμενη εβδομάδα αναφέρεται στην ανακοίνωσή σας για το 20% και περισσότερο και ενδεχομένω να αναφέρει το 30%. Γιατί το 20% δεν είναι προσφορά, δεν είναι κανένα είδου προσφορά, γιατί αυτό το έχουμε κάνει μονομερό. Άρα δεν είναι κάτι παραπάνω που προσφέρουμε. Θα πρέπει να υπάρχει ω σημείο πίεση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρχει κάτι παραπάνω σε δύο, σε τρία χρόνια. Παρακαλώ, ακούστηκαν πάρα πολλέ ερωτήσει. Ευχαριστώ πολύ και λυπούμε αν ε, δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες. Πρώτον, Ρίτσα Σίπερτ για το μοντέλο Primes. Δεν υπάρχει τίποτα καινούριο, χρησιμοποιείται για χρόνια και χρόνια. Το ενεργειακό τμήμα το έχει χρησιμοποιήσει η ειδική των χωρών μελών, το Euroelectrics, που είναι επίσης μια ένωση, το έχει χρησιμοποιήσει το μοντέλο αυτό και για το δικό της οδικό χάρτη του 2015. Συνεπώς δεν υπάρχει τίποτα το μυστηριώδης και όλα εξηγούνται στα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχει διαφάνεια δηλαδή. Μπορεί να ακούγονται διάφορα, αλλά δεν υπάρχει κανένα περίεργο, μυστικό, όπως ορισμένοι έχουν την τάση να πιστεύουν μερικές φορές. Για την ελαστικότητα τώρα των χωρών μελών και την ενεργειακή απόδοση. Ναι, φυσικά και πρέπει να υπάρχει κάποια ευελιξία και το προσπαθούμε. Προσπαθούμε να έχουμε ρυθμίσεις οι οποίες να έχουν προδιαγραφές η διάταξη για παράδειγμα γιατί να λέμε ότι έχουμε αποτύχει ενώ καταφέρουμε και κάνουμε πολλά όσον αφορά την κατασκευή των κτηριών. Είναι κάτι που δεν γίνεται στα κράτη-μέλη και αυτό είναι κάτι που καταστρέφει όλους μας εφόσον δεν εφαρμόζεται στα κράτη-μέλη. Και κάτι ακόμα. Ναι, ευελιξία. Αλλά όταν τώρα υπογραμμίζουμε τόσο πολύ μέσω της πρότασης της Επιτροπής για να στηρίξουμε τα κράτη-μέλη να κάνουν κάτι όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε και την αντίστοιχη συγκομιδή. Δεν μπορεί να κάνουμε την προσπάθεια να μην έχουμε τίποτα μετά. Είναι τα πιο καλά, αν συγκρίνουμε ε, την επένδυση και το κόστος, το καλύτερο μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας. Προκειμένου να πετύχουμε αυτή την απόδοση που θέλουμε. Λίντα, δεν ρώτησες κάτι, αλλά α, θα έχετε κάτι για την βιομάσα και τα κριτήρια βιωσιμότητας. Θα γίνει μια πρόταση πριν τα τέλη της χρονιάς από τον Επίτροπο Έτιγκερ. Ο Χρυκοκρόμα ρώτησε επίση για επιπλέον μέτρα, μέτρα αντιστοιχία δηλαδή, που προσπαθούμε να τα βρούμε με τις άλλες χώρες. Καταλαβαίνω, το παραδέχομαι. Αυτά που λέει ο τύπος δεν είναι πάντα τα σωστά. Έχουμε συζητήσεις για τις ισοτιμίες, τις αντιστοιχίε με άλλες χώρες. Με την Κίνα, για παράδειγμα, το έχουμε συζητήσει, με τη Ρωσία επίσης, το από την προηγούμενη εβδομάδα τον επόμενο μήνα επίσης θα υπάρχει μια συνάντηση ανάμεσα σε πυρογνώμονες Ρωσίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι δηλαδή κάτι που συζητιέται, τα ισοδύναμα. Και ήταν και μέρος της συνάντησης στο ΙΚΑΟ. Είπε η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορούμε να συζητήσουμε λίγο για τις ισοδυναμίες. Ρωτάτε κατά πόσο εξαιτία αυτή τη ιστορία με την αεροπορία θα πληγεί τον Τέρμπαν. Ειλικρινά δεν το πιστεύω. Σε όλου του άλλου τομεί, όλε οι άλλε χώρε ζητάνε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι πιο φιλόδοξη. Δεν θα ήταν περίεργο τώρα να λένε, μα δεν θα κάνετε κάτι με την αεροπορία. Ο, οι περισσότεροι θέλουν να γίνει. Εγώ καταλαβαίνω ότι θα ήταν καλύτερα να είχαμε μια συνολική ρύθμιση και το προσπαθούμε από το 1997. Τώρα προτείνουμε να συμπεριληφθεί η αεροπορία σαν ένας τομέας. Να μην είναι το βάρος μόνο στη βιομηχανία, στην ενέργεια, αλλά προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό με έναν τρόπο ο οποίος δεν θα πλήξει τους εταίρους μας, αλλά θα είναι κάτι λογικό και καλό για όλους. Και εκείνοι που εσείς μπορείτε να μας βοηθήσετε, να είναι σωστές οι αναλογίες. Γιατί μερικές φορές έχει κανείς την εντύπωση ότι όλες οι αεροπορικές εταιρείες θα αρχίσουν να πηγαίνουν στην Αποανατολή. Δεν ξέρω για σας, ξέρω για μένα και ξέρω για τους γνωστούς μου. Προκειμένου να κερδίσουν 2 ευρώ αν μπορούν να πάνε από το Πεκίνο στη Φραγκφούρτη για να κερδίσουν 2 ευρώ, δεν θα πάνε μέσω του Αμπουντάμπη και να περιμένουν 5-10 ώρες εκεί για να κερδίσουν 2 ευρώ. Υπάρχουν ε, ένα σώρο επιχειρήματα που ακούγονται που είναι εντελώς ανόητα. Και σε αυτό εσείς μπορείτε να βοηθήσετε στα κράτη-μέλη να περάσει το σωστό μήνυμα. 85% όλων ε, θα είναι δωρεάν τα πρώτα χρόνια. Τα τελμερικές φορές όταν ακούτε τα επιχειρήματα δεν μπορείτε να πιστέψετε ότι παίρνουν το 82,5% δωρεάν. Δεν νομίζω λοιπόν ότι εδώ θα υπάρξει καμία ζημιά στον Τέρμπαν. Και πάντα για την οπορία. Η ρώτησε Λέει γιατί δεν έχουμε συμμάχους. Έχουμε συμμάχους. Πάνω από 40 χώρες το κάνουμε. Έχουμε καλούς συμμάχους. Ο Καναδάς δεν υπέγραψε κατά της Ευρώπης του Αυστραλία. Κάνουμε πολλή δουλειά σε αυτό το τομέα. Χωρίς πάντως να μπούμε στις λεπτομέρειες, μπορείτε να καταλάβετε όλοι γιατί υπάρχουν μερικές μεγάλες χώρες που θέλουν να το καταπολεμήσουν και κάποιες αεροπορικές εταιρείε που θέλουν να τα καταπολεμήσουν. Αλλά προσοχή, οι αεροπορικές ε, εταιρείε ήταν κατά μια συνολική συμφωνία... και δεν έγινε. Τώρα προσπαθούν να μην περάσει ούτε και αυτό. Άρα κάτι τρέχει εδώ. Εγώ πιστεύω ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να υποκύψει σε εκβιασμούς και σε πιέσεις. Δεν θα δεχτούμε κάποιες χώρες να λένε αν καταργήσετε τη δικιά σας νομοθεσία, δεν την αλλάξετε, τότε εμείς θα έχουμε αντίπεινα. Όχι, πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Εγώ δεν ήμουν επίτροπος τότε, αλλά το Κοινοβούλιο ήξερε τι έκανε. Η Επιτροπή ήξερε τι έκανε. Και οι 27 χώρες μέλη ήξεραν τι έκαναν. Τίποτα δεν θα πρέπει να μας εκπλήσει εδώ. Αυτό πρέπει να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε να βρούμε καλές λύσεις στο τέλος. Ρωτήσατε επίση κατά πόσο θα είναι αρνητικό αν δεν πάρουμε μια δεύτερη περίοδο δεσμεύσεων. Όχι, θα έλεγα εγώ, σε σχέση με τις αναπτυσσόμενες χώρες. Πιστεύω ότι όπως είπαν ορισμένοι από εσά, δεν κάνει μεγάλη διαφορά για την Ευρώπη. Εμείς έχουμε τους στόχους μας είναι περασμένη στην νομοθεσία μας, είναι ξεκάθαρο το τι θα κάνουμε εμείς μέχρι το 2020. Είναι κακό όμως για τον κόσμο. Αν εμείς απλώς πούμε, εντάξει, εμείς θα πάρουμε μια δεύτερη περίοδο δεσμεύσεων, χωρίς προϋποθέσεις, θα το κάνουμε, τότε και πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι αυτή ήταν πάλι την άνοιξη που πολλές χώρες είπαν μόνο αν πάρει η δεύτερη περίοδο δεσμεύσεων, μόνο τότε θα είναι το τέρμαν μεγάλη επιτυχία. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι μεγάλο λάθος, γιατί αυτό δεν θα μειώσει κατά ένα παραπάνω τόνο τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και εγώ δεν βλέπω πώς μπορούμε να πούμε ότι είναι επιτυχία μια τέτοια διάσκεψη αν δεν υπάρχει προοπτική κάποιος να μπορεί να προσφέρει κάτι παραπάνω από αυτό που πρόσφερε μέχρι τότε. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να πούμε ότι ναι θέλουμε να αναλάβουμε αυτή την δεύτερη δέσμευση, Θέλουμε να κρατήσουμε ζωντανό αυτό που προσπαθήσαμε τόσο καιρό να φτιάξουμε και φτιάξαμε για το Κιώτο, αλλά για να φτιάξουμε το γεφύρωμα αυτό με το μέλλον είναι να δούμε ότι και άλλοι σε ένα βαθμό τουλάχιστον θα μας ακολουθήσουν. Το δεχόμαστε το ότι δεν πρόκειται να συμβεί αυτό παρέτα στον Τέρμπαν, αλλά πρέπει να ξέρουμε πότε και οι άλλοι θα ακολουθήσουν το δικό μας το παράδειγμα. Περί αυτού πρόκειται, αυτό είναι το Τέρμπαν. Και γι' αυτό και προσπαθούμε να πιέσουμε να πετύχει αυτό. Νομίζω ότι έτσι απαντά στον Φλόρενς. Α, βγήκε. Καλά. Εντάξει, θα είμαι πολύ σύντομη. Νομίζω... Ναι, θα έρθει. Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για μένα είναι ξεκάθαρα σε πολλούς τομείς. Εκεί που δεν είναι τόσο πολύ. είναι εκεί που θέλουμε να προσπαθήσουμε για το AUS να βρούμε κάποια, κάποιο συμβιβασμό. Ρωτήσατε επίσης για το EAS, την διπλωματία σε αυτό το επίπεδο. Τα κράτη-μέλη και πολλοί υπουργοί κάνουν πράγματα, αλλά για να συμπεριλάβουμε όλο, όλη την υπηρεσία εξωτερικής δράσης, είναι δύσκολο. Πολλές από τις αντιπροσωπείες μας ήδη κάνουν πολλή δουλειά και συνεργαζόμαστε μαζί τους έτσι ώστε να έχουν και αυτοί τα κατάλληλα επιχειρήματα, να ξέρουν που, πώς έχουν τα πράγματα στη διεθνή σκηνή και κάθε φορά που έχω την ευκαιρία πηγαίνω για να δω τι κάνουν. Ναι, μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα και να περιμένουν περισσότερο από αυτού, αλλά ήδη πολλοί από αυτού κάνουν εξαιρετικά πράγματα. Κύριε Σονούνη, δεν θέλω να μπω σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί εγώ δεν ξέρω την ιστορία αυτή με το εργοστάσιο στο Βένετο που μας είπατε. Πάντω αναφέρθηκα στη δεύτερη περίοδο δέσμευση. Αναφερθήκατε και στο IMO και τους δείχτες για τα πλοία. Πράγματι κάνει μια διαφορά όταν θα πρέπει όλα τα σκάφη να ναυπηγούνται βάσει των προδιαγραφών ενεργειακής απόδοσης, θα υπάρχει διαφορά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο τομέας δεν συνεχίζει να εκπέμπει όλο και, περισσότερες, ε, όλο και περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα. Γι' αυτό χρειάζονται και μέτρα στην αγορά. είτε κάποια εισφορά ανάλογα με τις εκπομπές, είτε εμπορία ε, εκπομπών και τα λοιπά, ανταλλαγές και τέτοια. Για τον Πιτελίζε, ρωτήσατε κάτι για τη διαρροή διοξιδίου του Άφρακα Αυτές είναι οι έμεσες εκπομπές. Εδώ η Γενική Διεύθυνση ΚΟΜ πολύ σύντομα θα έχει μία πρόταση πριν από τα τέλη της χρονιάς. Και ξέρω ότι είναι κάτι που συζητιέται πολύ στα κράτη-μέλη. Η κυρία Χάση τώρα ρώτησε για τη σχέση ανάμεσα στην εμπορία εκπομπών και τις πρωτοβουλίες για την ενεργειακή απόδοση. Στον οδικό χάρτη 2050 αναφέρεται μια σχέση. Πόσο δηλαδή σε aside πρέπει να έχεις και πόσοι... Ε, πόσες πρωτοβουλίες ενεργειακής απόδοσης. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε πάνω σε αυτό και ελπίζω κατά τη διάρκεια της Δανέζικης Προεδρίας να έχουμε καταλήξει που θα έχουμε και τον οδικό χάρτη για το χαμηλό άνθρακα και για το 2050 και την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση, οπότε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες θα μπορούμε να τις εξετάσουμε όλες μαζί συνολικά. Ε, με ρωτήσατε πότε θα πετύχει, με τι κριτήρια θα κρίνουμε ότι πέτυχε το Ντέρμπεν. Πρώτον, εφαρμογή όσων προβλέπονται να εφαρμοστούν μετά το Κανκούν. Είναι μεγάλος ο κατάλογος, αλλά είναι πολύ σημαντικό να έχουμε προχωρήσει εδώ πολύ. Δεύτερον, να προχωρήσουμε στο Πράσινο Ταμείο και τρίτον ο δικός χάρτης. Εσύ ρωτάτε κατά πόσο ο δικός χάρτης μπορεί να αντικαταστήσει την δεύτερη περίοδο δέσμευσης. Εγώ λέω ότι πρέπει να την πάρουμε αυτή την περίοδο, αλλά συγχρόνως να έχουμε και τον οδικό χάρτη και άλλα κριτήρια που να λένε ότι κάποια στιγμή και άλλες χώρες θα συμμετάσχουν. Περί αυτού πρόκειται. Όταν μιλάμε για τις αναδυόμενες οικονομίες, αυτό που θέλουμε είναι ένα νομικό παραλληλισμό. Δεν λέμε ότι άλλοι πρέπει να δεσμευτούν ακριβώς με τα ίδια νούμερα που δεσμευόμαστε κι εμεί. ούτε ζητάμε από τις αναδυόμενε οικονομίες να κάνουν τα πράγματα εξίσου φιλόδοξα, τόσο γρήγορα όσο θέλουμε να τα κάνουμε κι εμεί στις αναπτυγμένες χώρες. Λέμε όμως ότι ό,τι βάζουμε εμείς κάτι αναλογικά πρέπει να βάζουν και άλλοι στο μέλλον. Πρέπει να έχει όμως αυτό το οποίο υπόσχονται την ίδια νομική αξία. Αν εσείς βάζετε τόσα πολλά και οι άλλοι βάζουν πιο λίγα, μπορεί κάλλιστα να έχουν την ίδια νομική αξία. Μπορεί να μην είναι το ίδιο ποσό, αλλά σημαίνει πολλά αυτή η νομική βεβαιότητα. Πρέπει και εμείς να ξέρουμε ότι το αποτέλεσμα θα υπάρχει. Περί αυτού πρόκειται δηλαδή. Προς το παρόν χωρίζεται ο κόσμος, αλλά πόσο καιρό θα συνεχίσουμε με το παλιό καθεστώς και να θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα μείνουμε κάτω από 2%. Ανταυτού χρειαζόμαστε κάτι που να είναι περισσότερο προσαρμοσμένο στην πραγματικότητα. Δεν λέμε ότι θέλουμε οι άλλοι να αναλάβουν την ευθύνη, όχι, αλλά λέμε ότι τώρα στον 21ο αιώνα ό,τι προσφέρει ο καθένας πρέπει να έχει το ίδιο βάρος και να μετράει εξίσου. Και για να απαντήσω και στην αντιπροσωπεία του ΕΛΚ για το ποιο είναι ο ρόλος, πάντα έρχεται αυτό το θέμα και δεν πειράζει. Ξέρω η επόμενη ερώτηση θα είναι για τους 27 υπουργούς που εκπροσωπούν 27 χώρες και αυτοί έχουν τις δικές τους εθνικές επιτροπές, επειδή εσείς ζητήσατε να προσκληθεί ο δικός σας ο πρόεδρος. Και αυτοί θα ζητήσουν, οι δικοί τους οι πρόεδροι να προσκληθούν. Και αυτό είναι δύσκολο να το λύνουμε αυτό. Συνήθως έχουμε ένα καλό τρόπο και το λύνουμε. Έχουμε πολύ στενή συνεργασία και συντονισμό μεταξύ μας. Και να ξέρετε ότι εγώ θα είμαι στη διάθεσή σας και στη διάθεση του Προέδρου για ό,τι θέλετε. Τέλος. Ρωτάτε αν ε, εγώ πιστεύω ότι τα χρήματα θα τα έχουμε. Εγώ πιέζω το κράτη-mail και παρόλο που είναι δύσκολη η καιρή, ελπίζω ότι θα έχουμε τα χρήματα για το φάστα. Πιέζουμε. Η πίεση φέρνει αποτελέσματα Οπότε τις τελευταίες εβδομάδες συνεχίζουμε εν ώψη του Τέρμπαν και βλέπουμε ότι οι συνεισφορές των κρατών μελών αρχίζουν να φτάνουν. Συναντιέμαι και με χώρες, αφρικανικές χώρες ή άλλες που είναι Τώρα αρχίζουν και αντιλαμβάνονται ότι τα χρήματα αυτά από την Ευρώπη αρχίζουν να φτάνουν και ευχαριστούμε πολύ. Δεν είναι τέλεια τα πράγματα, αλλά αρχίζει να φαίνεται κάποια διαφορά. Ισραίουν τα χρήματα, αρχίζουν. Βέβαια, τα κράτη-μέλη πρέπει να φροντίσουν να φέρουν σε πέρα στις υποσχέσεις τους. Θα σας έκανε εντύπωση αν μαθαίνετε ποιες είναι οι χώρες οι οποίες ε, δεν δίνουν 100%. Πάντως και εσείς πρέπει να πιέσετε τις κυβερνήσεις σας για να προχωρήσουν. Ωραία. Υπάρχουν και κάποια άλλα ερωτήματα τα οποία θα απαντηθούν εν ευθέτω χρόνο. Uh, black, uh, ah, sorry, Yeah, ε, do we think, do I think Do I think that um, will help us? Για κατά πόσον πιστεύω ότι το αέριο από λιθό θα μας βοηθήσει να πετύχουμε τις φιλοδοξίες μας. Ρωτήσατε επίσης ε, αν η Ευρώπη σκοπεύει να κάνει μαζική επένδυση. Η απάντηση είναι αρνητική. Όχι σε αυτή τη φάση. Εξετάζουμε κατά πόσον όλη μας η νομοθεσία είναι εξοπλισμένη για να αντιμετωπίσει ενδεχόμενα προβλήματα που θα προκύψουν από το αέριο τους. Δεν το οργανώνουμε με την Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Ενεργείας κτλ. Με διαβουλέψεις με επιστήμονες, αλλά νομίζω ότι ο τρόπος που μπορούμε να φροντίσουμε να μην γίνουν σημαντικές επενδύσεις σε προβληματικά ζητήματα είναι να θέσουμε για το 2040 και το 2050 τα ορόσημα. Ευχαριστώ πολύ, ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε την Επίτροπο για την πολύ καλή αυτή παρουσίαση των ζητημάτων σε ό,τι αφορά τη δράση για το κλίμα. Νομίζω ότι καταλαβαίνουμε το τι κάνετε. Δεν ε, υπάρχει τελμάτωση. Θα τα πούμε είτε στο Στρασβούργο λοιπόν και στον Τέρμπαν καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας Γι' αυτό που ελπίζουμε ότι θα αποτελέσει μια επιτυχία για την COP17. Ευχαριστώ και τώρα στο 3G1 ε, θα συνδεθούν οι συντονιστές.